Okay, friends, we are not that many here yet, but we'll start with the first item on uh, the agenda for Λοιπόν, βλέπετε την ημερήσια διάταξη για σήμερα. Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Δημοκρατία της Κορέας θα δώσω το λόγο στον Σον Σάιμον. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Γι' αυτό το θέμα δεν υπάρχει πολύ πίεση χρόνου. Ίσως κάποιοι να θεωρούν ότι το θέμα είναι περιφοριακό νομικό, τεχνικό, δευτερεύον με λίγα λόγια. Παρ' όλα αυτά είναι νομίζω αρκετά σημαντικό θέμα. Δεν θα μακρηγορήσω, δεν θα σας κουράσω. Είναι ουσιαστικά η εμπορική συμφωνία που υπογράφηκε το 2011. Είναι η πρώτη συμφωνία από την λεγόμενη νέα γενιά, νέα σειρά συμφωνιών με ευνοϊκούς εμπορικούς όρους προς την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αλήθεια η συμφωνία επίσης ε, παρέχει πάρα πολλές ρήτρες, ε, προβλέπει πάρα πολλές ρήτρες και για την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων. Ως εκ τούτου είναι μια συμφωνία η οποία θα έπρεπε να μας ενδιαφέρει. Η γνωμοδότηση λοιπόν την οποία σας προτείνουμε, αν και είναι συνοπτική, έχει περιλαμβάνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα δηλαδή τα υψηλά επίπεδα προστασίας ε, των δικαιωμάτων των εργαζομένων είναι κάτι το οποίο δεν έχει γίνει σεβαστό από τους, ε, ε, από τους Κορεάτες από το 2011 μέχρι σήμερα. Έχουν υπάρξει επανειλημμένες διαμαρτυρίες από τα συνδικάτα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε εθνικά επίπεδα έχουν γίνει παραστάσεις διαμαρτυρίας προς τις πρεσβείες ε, της Δημοκρατίας της Κορέας. Η Κορέα συστηματικά αγνοεί συμφωνίες του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, δεν επικυρώνει τις συμφωνίες αυτές, παρεμποδίζει τις, τα συλλογικά δικαιώματα, τα δικαιώματα οργάνωσης, τα δικαιώματα διαμαρτυρίας με ε, συστηματικό και σοβαρότατο τρόπο. το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, η ομάδα των 10, ο ΟΣΑ, έχουν ε, προβλέψει ε, δύο, ε, έχουν μάλλον απαγορεύσει ουσιαστικά σε δύο επίπεδα κυρώσεις εις βάρος της Κορέας και η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της συμφωνίας αυτής έχει την δυνατότητα να πιέσει έντονα τους Κορεάτες για τον τρόπο με τον οποίο μεταχειρίζονται τους συνδικαλιστές και τα συνδικάτα στη χώρα τους. Αυτό το οποίο ζητάμε στη γνωμοδότηση της Επιτροπής μας, στην ουσία δηλαδή μια ενδιάμεση έκθεση, είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρακολουθήσει από κοντά εκ του σύνεγγες λοιπόν τις συγκεκριμένες εξελίξεις στη δημοκρατία της Κορέας. Δεν είναι υπερβολικό το αίτημα αυτό, ιδιαίτερα για την δική μας Επιτροπή, την Επιτροπή Απασχόλησης, σε έναν τομέα ο οποίος κυρίως θα έλεγα έχει σημασία γιατί όπως είπα η εμπορική συμφωνία είναι μια νέα γενιά συμφωνιών. Λοιπόν αυτό είναι η ουσία, έχει σημασία η συμφωνία αυτή εγώ δεν προβλέπω να υπάρξει ένα πάρα πολύ ε, χρονοβόρο ε, διάστημα. Τροπολογίες στις 29 Απριλίου θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας ε, στις 15 ή 16 Ιουνίου. Ελπίζω να μην έχουμε πάρα πολλές τροπολογίες, να μην είναι πολύ δύσκολες και να μπορέσουμε γρήγορα να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία από όλες πλευρές. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Δεν είναι εδώ ο σκιώδης του Ελκ. Ούτε η Γκέρι και είναι εδώ. Ίσως η Χέλγκα Στίβενς να ήθελε το λόγο. Θα έλθει αργότερα. Από την ομάδα των φιλελευθέρων. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συνάδελφοι, θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την πρόταση γνωμοδότηση την οποία κατέθεσε. Η Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών Ένωσης Κορέας είναι καινοτόμα στον τομέα των εμπορικών σχέσεων και της αηφόρου ανάπτυξης καθώς το, και στο θέμα του περιβάλλοντος και των εργασιακών σχέσεων. Θα πρέπει λοιπόν να τηρούνται οι προδιαγραφέ του Διεθνού Οργάνωση Εργασία, συμπεριλαμβανομένων και τα βασικά δικαιώματα των εργαζομένων και βέβαια να τηρηθεί η δέσμευση για την υπογραφή και κύρωση όλων των συμβάσεων τη Διεθνού Οργάνωση Εργασία. Νότια Κορέα δεν έχει ακόμα κυρώσει κύριες Τέτοιε συμβάσει όπω τη σχετική με την ελευθερία του τη, δεν σε την ουσιαστική αναγνώριση του δικαιώματο τη λογική διαπραγματεύση και τον προσδιορισμό τη καταναγκαστική εργασία. Απευθύνεται έκκληση λοιπόν στην Νότια Κορέα να επιταχύνει την κύρωση των συμβάσεων αυτών και ταυτόχρονα πρέπει να αναγνωριστεί ως σημαντικό βήμα το γεγονός ότι έχουν συμφωνήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Κορέα την ε, κύρωση της ε, σύμβασης του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας για την αποφυγή διακρίσεων ως προς τα δικαιώματα των εργαζομένων. Έτσι μπορούν να εξασφαλίζονται αυτά με ένα στενότερο διάλογο μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Νότιας Κορέας στο πλαίσιο των προβλεπωμένων στη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών. Το πνεύμα λοιπόν που προκύπτει πρέπει να προχωρεί με βάση τις προδιαγραφές, τις ύψες προδιαγραφές για τις συνθήκες εργασίας και αυτή πρέπει να είναι η κατεύθυνση που θα ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Νότια Κορέα. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Άρη Ρόνια Κάρη, Σας ευχαριστώ. Θα <clears throat> μιλήσω δανεικά, επομένως σας καλώ να φορέσετε ακουστικά, λέει ο Μιλήτρια. Πρώτα απ' όλα να πω ότι συμφωνώ ότι πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό θέμα. Έχουμε την συγκεκριμένη πρόταση επιτάπητος, αλλά έχουμε και ένα γενικότερο θέμα προσέγγισης τέτοιων συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών με χώρες που χειρίζονται έτσι τα εργασιακά του ζητήματα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ για το σχέδιο. Έχει πάρα πολλά καλά στοιχεία παρά το σύντομο του κειμένου. Θα ήθελα να ενισχύσουμε ορισμένα σημεία, να υπογραμμίζουμε τα θέματα παραβιάσεων δικαιωμάτων, αλλά να υπογραμμίσουμε και το γεγονό ότι θα υπάρχουν συνέπειε αν η Κορέα δεν εγγυηθεί τα θεμελιώδη δικαιώματα των εργαζομένων. Δεν μπορούμε να έχουμε FTAs χωρίς να υλοποιούνται, να εφαρμόζονται, να τηρούνται όλα τα δικαιώματα του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας. Πρέπει λοιπόν να υπογραμμίσουμε το γεγονός ότι αν συνεχίσουν έτσι, οι Κορεάτες θα υπάρξουν συνεπείς. Κατά τα άλλα σύμφωνο. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μέσεριτς είναι εδώ από τους Πρασίνους. Όχι και δεν βλέπω να υπάρχει και αντικαταστάτης. Τιτσιάνα Μπέγκιν, η παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλημέρα, συνάδελφοι. Να ευχαριστήσω και εγώ τον εισηγητή για, ένα, για μια πολύ καλή δουλειά. Και εγώ συμφωνώ ότι οι συμφωνίε ελευθέρων συναλλαγών που υπογράφουμε με τους εταίρους μας θα πρέπει να είναι και εργαλεία προώθησης των θεμελιωδών αξιών μας και αρχών. Στην πραγματικότητα εδώ αυξάνεται η ένταση και η αντιπαράθεση μεταξύ της κυβέρνησης και των ενώσεων των εργαζομένων. Συμφωνώ με τις, ε, με τις επισημείωσεις που έχουν γίνει για τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων, αλλά θυμίζω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνουμε αυτό, παρά τις ρήτρες προστασίες που προβλέπουν οι συμβάσεις και οι συνθήκες. Όταν λοιπόν έχουμε διευκολύνσεις εμπορικές, είτε έχουμε ε, συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών, η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε θέση ισχύω για να πιέζει για αυτά τα ζητήματα. Η Κορέα πιο συγκεκριμένα είναι πάρα πολύ σημαντικό να επικυρώσει όλες τις συμφωνίες υπό τον ILO, όπως και τις καταναγκαστικές εργασίες. Η Νότια Κορέα εποφελήθηκε από τη συμφωνία αυτή έντονα από τους όγκους ε, συναλλαγών και επομένως τώρα καλό θα είναι να προστατεύσει και τον πληθυσμό του και τους εργαζομένους της. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η Μάρα Μπιζότ ε, δεν είναι εδώ. Ο κύριος Ντομινίκ Ματά. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Ε, συγχωρήστε την ε, κυρία Μπιζότο η οποία είχε άλλα, άλλες υποχρεώσεις να σας πω με εδώ λέω για την απόψή μου καταρχάς να συγχαρώ τον εισηγητή έχουμε την εντύπωση ότι πρόκειται για μια ανταλλαγή ναι θα κάνουμε εμπόριο μαζί σας εφόσον δεσμευτείτε ότι θα σεβαστείτε τα θεμελιώδη δικαιώματα του ΑΕΛΟ αυτή η ανταλλαγή μου φαίνεται λίγο περιπετειώδης και αμφίβολη. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι η Νότια Κορέα με τις συνήθειες που έχει ήδη αναπτύξει τελικό θα τηρήσει αυτές τις υποχρεώσεις. Ιδιαίτερα σε σχέση με την αναγκαστική εργασία. Και για τη δήλωση της κυρία Βυζότου σας διαβάζω. Η εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρόκειται, αντιπροσωπεύει ένα κίνδυνο και απειλή ιδιαίτερα για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μας που εργάζονται ε, στον τομέα της ε, περιφερειακής αριστείας και υψηλής ποιότητας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σε πάρα πολλούς οικονομικούς τομείς πολύ σημαντικούς έχει, δεν έχει προστατεύσει τη στρέβλωση της ανταγωνιστικότητας μεταξύ των χωρών και των περιφερειών και αναφέρομαι ιδιαίτερα στις γεωγραφικές ενδείξεις προέλευσης και παραδοσιακά προϊόντα όπως τα ελλαντικά, το τυρί κτλ. Εξακολουθούμε να υπογράφουμε συμφωνίες που παραβιάζουν κατάφορα τα δικαιώματα των παραγωγών μας. Έχουμε μπροστά μας μια συμφωνία ελευθερών συναλλαγών με το Βιετνάμ όπου μετατρέπουμε τις ε, γεωγραφικές ε, ονομασίες προέλευσης ως ε, τυπικό, τυπική ονομασία. Δηλαδή θα μπορούμε να έχουμε καμομπέρ, το οποίο θα παρασκευάζεται στην Αλαμπάμα. Και έτσι, στην ουσία, παρακάμπτουμε την πραγματική προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων. Πρέπει περιοδικά και συστηματικά να επανεξετάζουμε όλες τις συμφωνίες που υπογράφουμε και τον αντίκτυπό τους για όλους τους τομείς της οικονομίας, ώστε να μπορούμε να έχουμε κυρώσεις τελωνιακές σε περίπτωση παραβιάσεων. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών με την Κορέα είναι ένα θετικό βήμα και το σχέδιο γνωμοδότησης είναι στη σωστή κατεύθυνση. Από την πλευρά μας, σαν Επιτροπή Απασχόλησης, πρέπει να επιμείνουμε έτσι ώστε, εκτός από το σεβασμό των εργασιακών δικαιωμάτων, να εστιάσουμε στο γεγονός ότι στην Κορέα η παιδική εργασία είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα. Επίσης, η ασφάλεια στην εργασία είναι ένα άλλο σημαντικό θέμα το οποίο πρέπει να κοιτάξουμε. Δυστυχώ, στη χώρα που δραστηριοποιούνται πολυεθνικές πάρα πολλές πολυεθνικές, θεωρώ αμφίβολη αν μπορούμε να τους αλλάξουμε την νοοτροπία που μπροστά στο κέρδος δεν σέβονται τίποτα. Σας ευχαριστώ. Thank you. Uh, we have Ευχαριστώ. Έχουμε εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου. Θα σας δώσουμε και τη δική μας άποψη. Αυτή η συμφωνία με την Κορέα λοιπόν εφαρμόζεται τώρα, βρίσκεται στον πέμπτο χρόνο, έχουν εφαρμοστεί τα περισσότερα κεφάλαια κατά τη διάρκεια αυτών των τεσσάρων ετών συνεργαζόμεθα, υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη με τους Κορεάτες, έχουμε προχωρήσει σε μια λειτουργική ευρυθμία θα έλεγα μαζί τους. Έχουμε επίσης οργανώσει πολλές συναντήσεις και σε επίπεδο κοινωνίας των πολιτών. Εμείς ενημερώσαμε τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών για τις συναντήσεις μας με την κυβέρνηση της Κορέας και έχουμε δημοσιεύσει και κοινά ανακοινωθέν σχετικά με τις συζητήσεις μας η οποία ε, δεν ήταν κάτι το υποχρεωτικό να γίνει. Τώρα, σχετικά με τις επιμέρους συζητήσεις, νομίζω ότι τα θέματα είναι πολλά και ενδιαφέροντα. Τα βασικά θέματα είναι η επικύρηση των τεσσάρων βασικών θεμελιωδών συμβάσεων του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας που δεν έχει επικυρώσει η χώρα αυτή ακόμα έχει αναλάβει την υποχρέωση ε, να προχωρήσει στη διαδικασία επικύρωσης. Επίσης για την ε, θεμελιώδη σύμβαση 1.1.1 για την έλλειψη διακρίσεων στον τομέα της απασχόλησης και εργασίας. Και υπάρχει και το θέμα που έχουμε συζητήσει της αντιμετώπισης των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Εμείς είμαστε γενικά ικανοποιημένοι από τον τρόπο με τον οποίο συζητάμε τα θέματα αυτά με τους Κορεάτες. Νομίζω ότι οικοδομούμε μια επικοδομητική λύση ε, με την Κορέα και δεν χρειάζεται στην παρούσα φάση περαιτέρω δράση. Νομίζω ότι σε επίπεδο επιτευγμάτων να μου επιτρέψετε να σημειώσω ότι ξεπεράσαμε την διστακτικότητα της Κορέας να συζητήσει τα θέματα αυτά. Τώρα τα συζητάμε και πολλές φορές πολύ ανοιχτά και επιθετικά. Ε, η Κορέα επίσης ε, έχει δεχθεί τη συμμετοχή των εμπειρογνωμόνων του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας στις διακυβερνητικές συναντήσεις, κάτι το οποίο δεν ήταν δεδομένο στο παρελθόν λόγω των δύσκολων σχέσεων που είχε η χώρα αυτή με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας. Η Κορέα έχει επίσης ε, κάνει κάποια πρώτα βήματα για την επικύρωση των τριών συμβάσεων, κάτι το οποίο δεν έχει ολοκληρώσει και τέταρτον έχει δημιουργηθεί η πλατφόρμα για την επαφή των συνδικάτων και των ε, ε, εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών και έτσι έχουμε την δυνατότητα να θέσουμε τα θέματα αυτά άμεσα προς την κυβέρνηση της Κορέας. Νομίζω ότι δεν είχαμε μέχρι τώρα πλαίσιο για να το κάνουμε. Πέμπτον, Ξεκινάμε τις επόμενες μέρες με ένα νέο πρόγραμμα στα πλαίσια της εταιρικής σχέσης, του εταιρικού μέσου, για την αναθεώρηση της, του σεβασμού, αν θέλετε, της, της Σύμβασης 1-1-1 του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Προσπαθούμε να εντοπίσουμε τις βέλτιστες πρακτικές ε, για να δούμε ακριβώς ε, τι κάνει στον τομέα αυτό η Κορέα, αλλά όχι μόνον αυτή. Η διάσταση αυτή φυσικά θα αντιμετωπιστεί και στα πλαίσια της αξιολόγησης της εμπορικής συμφωνίας, η οποία θα ξεκινήσει το συντομότερο. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό ήταν ένα από τα δύο, ήταν μία από τις δύο πιο συζητημένες εμπορικές συμφωνίες, τις οποίες ξεκινήσαμε να συζητάμε από την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο. Το ένα ήταν η Κολομβία, το άλλο είναι η Κορέα. Έχει πολύ ενδιαφέρον θα έλεγα να προχωρήσει κανείς σε περαιτέρω συζητήσει και αξιολογήσεις. Θα ξαναδώσω το λόγο στο Σάιμον για να κλείσει το θέμα. Thank you very much. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους και οδησυγητές, μεταξύ των οποίων καταγράφω ευρεία συνένεση. και ελπίζω ότι μπορούμε να έχουμε μια συνεργατική διαδικασία, ταχεία διαδικασία. Βλέπω μία μόνο απόκληση από το σχέδιο της έκθεσης με την επιθυμία από κάποιους συναδέλφους να ζητήσουμε περισσότερα με πιο σαφή ορολογία και αναφορά σε κυρώσεις. Νομίζω ότι ο λόγος για τον οποίο το αποφύγαμε αυτό, δεδομένου ήταν το γεγονός ότι ξέρουμε πως πρόκειται για γνωμοδότηση μόνο της Επιτροπής ε, Απασχόλησης. Και ξέρουμε ότι η Επιτροπή Ίντρα που έχει, Ίντα που έχει την ε, κύρια έκθεση θα προσανατολιστεί περισσότερο προς τις πτυχές διεθνούς εμπορίου και τα σχετικά συμφέροντα. Γι' αυτό θέλησαμε να είμαστε πιο ρεαλιστικοί, πιο μετρημένοι. Βεβαίως, στην απάντηση της Επιτροπής Βλέπουμε τα στοιχεία αυτά και θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ την Επιτροπή για την εξαίρετη γραφειοκρατική ορολογία που χρησιμοποιεί σε ορισμένα σημεία στην υπενθύμηση της δέσμευσης της συμφωνίας για μια διαδικασία ε, κυρώσεων και όχι κυρώσεων ε, ε, αυτών καθεαυτών, όχι γυμνών κυρώσεων, πράγμα το έχει τεράστια σημασία και ιδιαίτερα το γεγονό ότι εν γέννη αισθάνεται ικανοποιημένη η Επιτροπή ε, με τις ε, προόδους στο χώρο των, εργασιακών, ε, των εργασιακών συνθήκων. Πέντε χρόνια που υπάρχει αυτή η συμφωνία το να ξυλοκοπούνται οι συνδικαλιστές και να ρίχνονται στη φυλακή δεν είναι ακριβώς η αντίληψη της θετικής εξέλιξης, αλλά μάλλον η απουσία πρόοδου. Πάντως, όταν υπάρχει δέσμευση για κύρωση και δέσμευση για ένταξη σε μια διαδικασία κυρώσεως των συνθήκων του Διεθνούς Οργανισμού, είναι κάτι διαφορετικό από την δέσμευση βεβαίως και αυτό πάλι ε, θα πρέπει να μας, ε, να μας κάνει ότι ξυλοκοπούνται και έρχονται στη φυλακή οι συνδικαλιστές. Και εγώ νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και εντό εισαγωγικών το βάζω, θα αισθανθεί γενικώ ικανοποιημένο από την πρόοδο των ε, ε, διαπραγματεύσεων. Ίσως λοιπόν θα πρέπει ως Επιτροπή Απασχόληση να μας απασχολήσουν και οι προτάσεις των συναδέλφων που θερούν πιο σκληρή γλώσσα και διεκδικούν περισσότερα. Γιατί μετά από αυτά που άκουσα από την Επιτροπή, πολύ φοβούμαι ότι θα εξασφαλίσουμε λιγότερα και από αυτά που θέλουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Όπως αναφέρατε και εσείς ξεκινώντας κύριε Σάιμον. Προθεσμία 28 Απριλίου. 15 ή 16 Ιουνίου η έγκριση στην Επιτροπή μας. Για την Ολομέλεια δεν έχουμε ιδέα. Και σας ευχαριστώ. Έχουμε πολλά θέματα Διεθνούς Εμπορίου στην Επιτροπή μας. Τελευταίος. φυσικολογικό μου φαίνεται. Σημείο 9 στην Εμερήσια διάταξη. Και πάλι οδηγία για, την, ε, για τις ότιμες συνθήκες απασχόλησης. Το έχουμε ξαναδεί. 310 τροπολογίες είχαν κατατεθεί και παρακαλώ την συγκεκριμένη να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που υπέβαλαν τροπολογίες γιατί είναι ένα από τα ευτυχή στοιχεία του οίκου μας Όταν δηλαδή οι τροπολογίες κινούνται προς αντίστοιχη κατεύθυνση και δεν έχουμε έντονα αποκλίνουσες. Κάποιες από τις τροπολογίες ζητούν μια διαφορετική απόχρωση ή ένα διαφορετικό τονισμό, αλλά συνολικά θεωρώ ότι έχουμε μια ομοιογενή προσέγγιση σχετικά με το πώς θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε τις διακρίσεις στο χώρο της εργασίας. Σχετικά με τις διακρίσεις τις ηλικιακέ. Νομίζω ότι εδώ υπάρχει στην ουσία ομοφωνία ότι και οι νέοι και οι ηλικιωμένοι θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και κατάλληλες πολιτικές θα πρέπει να εφαρμόζονται για την καταπολέμηση αυτών των διακρίσεων. Για τους άνω των 50 ετών η διαβίου μάθηση είναι η σωστή στάση όπως και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων πληροφορικής, ώστε να μπορεί κανείς να ανταπεξέλθει στις απαιτήσει της σημερινής ζωής και της σημερινής αγοράς κυρίως. Θα έλεγα ότι οι περισσότερες τροπολογίες αφορούν στην δική μας κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την ενσωμάτωση και την ένταξη των μεταναστών και την ανάγκη της σωστής ένταξής τους εις, την, τον κόσμο της εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τις αναπηρίες και χαίρομαι που και η κυρία Στίβενς είναι εδώ ακούσαμε, είδαμε την έκθεση ε, σχετικά με την υλοποίηση της σύμβασης για τους ανθρώπους με ανεπηρίες. Μερικές από τις ορπολογίες που υπέβαλε η κυρία Στίβενς είναι στην πραγματικότητα τα ουσιαστικά στοιχεία της έκθεσης εκείνης. Αρκετές από τις τροπολογίες υπογραμμίζουν ότι η έλλειψη ασφάλισης και η έλλειψη κατάλληλης κατοικίας σε αρκετές περιπτώσεις είναι στον καρδιά του προβλήματος. Συζητήσαμε και πολλές συμβιβαστικέ τροπολογίες για να μπορέσουμε να μειώσουμε λίγο τον αριθμό. Θα έχουμε 30 συμβιβαστικέ που ελπίζω ότι θα βελτιώσουν την έκθεση θα αφαιρέσουν κάποιες επικαλύψεις και θα την κάνουν πιο ευανάγνωστη στις συμβαστικές ενσωματώσαμε και κάποια πράγματα που έχουν ήδη ψηφιστεί στη ΛΥΜΠΕ και στην Φά διότι και αυτά συνάδουν προς τη γενική κατεύθυνση της γνωμοδότησης. Και πραγματικά επαναλαμβάνω ότι είναι ευτυχές ότι συμφωνούμε σε αυτά τα ζητήματα, από ό,τι φαίνεται όλοι, θα αποσταλούν αυτές εις τους σκιώδεις σήμερα πριν το μεσημέρι κατά τη και προβλέπεται μια συνάντηση για τους κοιόδης αύριο, αλλά μάλλον θα ήταν καλύτερα αυτό να γίνει την Πέμπτη, ώστε να εξεταστούν, να υπάρξει χρόνος για την εξέταση των συμβαστικών, αλλά αυτά είναι λεπτομέρειες. Που θα τις διαθετήσουμε μετά τη συνάντηση. Να ευχαριστήσω λοιπόν όλους τους συναδέλφους για τη συνεργασία και ελπίζω τελικά να έχουμε μια εύρωστη και σωστή γνωμοδότηση που θα μας βοηθήσει όλους στο μέλλον στη δουλειά αυτή. Σας ευχαριστώ. Θα δώσουμε τώρα το λόγο στους σκιώδεις. Η κυρία Ζάγεβιτς, παρακαλώ. Ε, dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo. Ε, przede wszystkim Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, συγχαρητήρια στη συντάκτρια. Πρόκειται για ένα σημαντικό θέμα, σημαντικό για μας και όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι προσλαμβάνει όλο και μεγαλύτερη σημασία και λόγω της μεταναστευτικής κρίσης και της νέας κατάστασης στην Ευρώπη ως προς την αντίληψη της ιδέας της αποφυγής των διακρίσεων και μέσα από τα όσα ορίζει η οδηγία ως παράγοντες ε, θρησκεία, αναπηρία ε, και άλλα. Με τη θρησκεία όμως σε πρώτη θέση. Είναι σημαντικό λοιπόν αυτό και αξίζει τον κόπο να το συστήσουμε. Και μια και είναι τόσο άμεση συνάφεια της οδηγίας, με όλη την εγκύτητα στις απόψεις θα πρότεινα να ματαιωθεί η συνεδρία των σκιωδών συντονιστών, γιατί χρειάζεται να ε, έχουμε προς να μελετήσουμε τις συμβαστικές τροπολογίες. Εάν ζητούμε σε άλλα έγγραφα ένα πιο ισορροπημένο τρόπο εργασία, δεν θα πρέπει να επιβάλλουμε στου δικού μα συνεργάτε εντατικού ρυθμού δουλειά που δεν θέλουμε για του υπόλοιπου εργαζομένου. Νομίζω ότι χρειάζεται λίγο πιστρο χρόνο. Ίσως για Τετάρτη. Για τη διαδικασία την ίδια τώρα. Ε, στο κείμενο βλέπω αρκετές επαναλήψεις σε σχέση με την ηλικία και την αναπηρία. Επίσης, ε, θα μπορούσαμε να προτείνουμε μια νέα αντίληψη με την παραπομπή στην ε, συνθήκη, στη Σύμβαση των Ηνωμένων για την Αναπηρία και επίσης η αναπηρία σχετίζεται με το περιβάλλον. Εάν ε, το περιβάλλον, ο χώρος, η κοινωνία είναι σχεδιασμένη κατάλληλα, δεν υπάρχουν φραγμοί λόγω αναπηρίας. Φερρυπίν φοράμε γυαλιά, έτσι. Πολλοί είναι αυτοί που φοράνε γυαλιά. Εάν όμως οι συνθήκες ε, των, ε, ε, του περιβάλλοντος που δεν μπορούσε κανείς να έχει τα γυαλιά του, δεν θα μπορούσε να βλέπει τίποτα, άρα θα ήταν καταδικασμένος σε έναν αποκλεισμό. Ε, το ίδιο λοιπόν χρειάζεται για όλους. Ο σχεδιασμός λοιπόν έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και ως τροπολογία θα έχει τεράστια αξία ώστε να πείσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να υποστηρίξουμε το, τα κράτη-μέλη να καταστήσουν πιο ευρέως δεδομένες τις δυνατότητες αυτές. να ενθαρρυνθούν ε, τα κράτη-μέλη ώστε να γίνει πιο δεδομένη η χρήση αυτών των δυνατοτήτων. Ε, αν εντατικοποιηθεί η προσπάθεια, η ευρωπαϊκή μπορούμε να φέρουμε καλύτερες λύσεις. Τροπολογίες σημαντικές υπάρχουν και για την, λειτουργία, για την συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασία ε, δεύτερη πρόσβαση, γιατί υπάρχουν πολλά ζητήματα σε επίπεδο κρατών μελών που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασία. Ωστόσο, μερικέ φορέ αυτέ οι διατάξει έχουν να κάνουν με ειδικέ μορφέ απασχόληση, ειδικέ συνθήκε. Έτσι λοιπόν ο καλύτερος τρόπος είναι να προσφέρουμε στους εργοδότες εργαλεία που θα εξασφαλίζουν για το άτομο με αναπηρία τελικά καλύτερη ευκαιρία πρόσβασης στην αγορά εργασίας για να διευκολυνθεί και η ενσωμάτωσή τους και να ενισχυθούν οι σχέσεις τους με τους λοιπούς εργαζομένους. Εάν ένα άτομο με αναπηρία εργάζεται σε κανονικές συνθήκες στην αγορά εργασίας και όχι σε ειδικέ συνθήκες, γιατί χωρίς να είναι γκέτο αυτές δεν διευκολύνουν ε, την ενσωμάτωση, νομίζω ότι θα έχουμε πολλά ε, θετικά. Η ψηφιοποίηση της αγοράς επίσης έχει τεράστια σημασία γιατί αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμεθα, αλλάζει την οργάνωση της εργασίας και ενώ κάποιοι την αντιλαμβάνονται αυτήν ως απειλή, εμείς κατά κύριο λόγο τη βλέπουμε ως ευκαιρία και ιδιαίτερα για όσους έχουν προβλήματα σε σχέση με την κινητικότητα. Νέες λοιπόν μορφές απασχόλησης που εξασφαλίζει η ψηφιοποίηση θα έχουν ιδιαίτερα, θα έχουν ιδιαίτερα ωφέλη να προσφέρουν στα άτομα με αναπηρία ή στους ε, πιο ηλικιωμένου. Για την αποφυγή των διακρίσεων των σχετικών με την θρησκεία επίσης. Με χαρά σημειώνω πως στην έκθεση υπάρχει αναφορά στο πεδίο εφαρμογή της οδηγίας καθώς η περίπτωση σύγκρουση συμφερόντων παραμένουν ενισχύει οι εθνικές διατάξεις. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Διότι ενώ ζητούμε πιο ουσιαστική αποφυγή των διακρίσεων ή αποτροπή των διακρίσεων, λησμονούμε συχνά στην περίπτωση των θρησκευτικών μειονοτήτων ότι πρέπει και οι δύο πλευρές να ισορροπούν ως προς το ευρωπαϊκό συμφέρον. Και αν δεν υπάρξει αυτή η ισορροπία δεν θα είναι καλή η έκθεση. Κύριε Βίλκεβισούτε, σκιώδης του Σοσιαλιστών. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την εισηγήτριά μας γιατί δείχνει ότι κατανοεί το ότι θα πρέπει να υπάρξει στενή συνεργασία μεταξύ μας και αναζήτηση συμβιβαστικών προτάσεων. Η πρόταση την οποία κάνει είναι πάρα πολύ καλή και μας δίνει την δυνατότητα να ξεπεραστούν κάποια από τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στις χώρες μέλη. Εμείς έχουμε καταθέσει σαν πολιτική ομάδα αρκετές τροπολογίες οι οποίες αντικατοπτρίζουν τις ανησυχίες μας. Το θέμα της ηλικίας καταρχάς είναι σημαντικό για μας. Λόγω των δημογραφικών αλλαγών στην Ελλάδα, λόγω της παράτασης της ηλικίας συνταξιοδότησης, οι διακρίσεις με βάση την ηλικία είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό και εφόσον από τη μία λαμβάνουμε αποφάσεις για την παράταση της εργασιακής ζωής, θα πρέπει να δώσουμε την δυνατότητα στους ηλικιωμένους πολίτες να παραμένουν στην αγορά εργασίας και να συμμετέχουν πλήρως σε αυτή. Θέλουμε λοιπόν να ενισχύσουμε την προστασία για ενάντια στις άδικες απολύσεις, να γίνονται σεβαστά τα όρια συνταξιοδότησης, και να αναλυθεί από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής το πρόβλημα της ε, ανεργίας των ε, συμπολιτών μας άνω των 50 ετών. Θα πρέπει να μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να επανέρχονται στην αγορά εργασίας και να επανεντάσσονται στην εργασία. Δεν πρέπει να υπάρξει αντιπαράθεση ανάμεσα στους νεότερους και τους παλαιότερους και οι διαφορετικές γενιές πρέπει να εκμεταλλεύονται την εμπειρία ημέν των δε. Απαιτείται καλύτερη συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους. Πρέπει να ενθαρρύνουμε επίσης και την διαβίου κατάρτιση. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να δείχνει ότι σεβόμεθα όλες τις κατηγορίες ηλικιών των εργαζομένων και θα πρέπει να είναι ε, τα προγράμματα κατάρτισης ανοιχτά σε όλους και για όλους. Πέρα από το θέμα της ηλικία έχουμε το θέμα της αναπηρίας. Δυστυχώς στην παρούσα φάση δεν είμαστε σε θέση να προστατεύσουμε από τις διακρίσεις τους ευάλωτους αυτούς ανθρώπους. Ορισμένες χώρες δεν εφαρμόζουν αυτή την πλευρά της οδηγίας, διότι δεν είναι σε θέση να προσαρμόσουν κάποιες θέσεις εργασίας ε, στις ανάγκες των αναπήρων και δεν παρέχουν όλες τις δυνατότητες κατάρτισης και εκπαίδευσης τους ανάπηρους. Πρέπει λοιπόν τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν ορθότερα τα διαρθρωτικά ταμεία για να υπάρξουν δυνατότητες απασχόλησης και για τους ανθρώπους με αναπηρία. Οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Και έτσι μόνο θα καταπολεμήσουμε τον κοινωνικό αποκλεισμό και τη φτώχεια. Ένα τρίτο θέμα είναι το θέμα των προβλημάτων στην, στο χώρο εργασίας, στο χώρο απασχόλησης. Ε, το θέμα της παρενόχλησης του χώρο εργασίας. Το ασπέκτο ε, darbo aplinkoj. Να, ir kartu turim pabrėžti, kad... Πρέπει λοιπόν να διαυκρινίσουμε ότι οι διακρίσεις εις βάρος των εργαζομένων πολλές φορές, ακόμα και για έμπειρους εργαζομένους, είναι κάτι για το οποίο δεν μπορεί να διαμαρτυρηθούν εύκολα οι εργαζόμενοι, φοβούνται να το κάνουν γιατί θα χάσουν τη δουλειά τους. Και επίσης πάρα πολλοί εργαζόμενοι δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και γι' αυτό και πρότεινα μία τροπολογία στα πλαίσια των επαφών με τις οργανώσεις των κοινωνικών εταίρων να υπογραμμιστεί το πρόβλημα του εκφοβισμού λοιπόν και της παρενόχλησης και πώς μπορεί το θέμα αυτό να ληφθεί υπόψη και στα πλαίσια των συλλογικών διαπραγματεύσεων και στα πλαίσια των επαφών ανάμεσα στην εργοδοσία και τους εργαζομένους. Θα πρέπει λοιπόν οι κοινωνικοί εταίροι, οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, η κοινωνία των πολιτών να έχει λόγο στα πλαίσια των ετοιμάτων για ισότιμη μεταχείριση των εργαζομένων. Και θα πρέπει τα κράτη-μέλη να ανταλλάξουν τις ε, καλές εμπειρίες που έχουν. Είμαι σίγουρη ότι θα καταλήξουμε σε κάποια συμβιβαστική λύση Ίσως η συνάντηση την Πέμπτη να είναι χρήσιμη. Στίβενς, έχετε το λόγο από τους συντηρητικούς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω όλους ε, τους ε, συναδέλφους. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα για το τμήμα της νομοδότησης ε, για τους ανθρώπους με αναπηρίες, όπως και τις καταληκτικές τους ε, παρατηρήσεις. Για τον εισηγητή και τη Λίμπε θα ήθελα να πω ότι οι διακρίσεις ε, ή μάλλον η αντιμετώπιση των διακρίσεων στον χώρο της εργασίας μπορούν να είναι αποτελεσματικές μόνο όταν συνοδεύονται σε όλη την προσωπική ζωή του ανθρώπου. Επομένως, τα... θα πρέπει να υπογραμμίσουμε τα δικαιώματα στην εργασία τα δικαιώματα στην κατάλληλη, στην κατάλληλη στέγαση σε συνδυασμό με την ε, ελεύθερη μετακίνηση και το δικαίωμα στην ελεύθερη μετακίνηση των ανθρώπων με αναπηρία. Για τους ανθρώπους άνω των 50 θα έπρεπε επίσης να υπογραμμίσουμε κάπως περισσότερο το πρόβλημα της εξέβρεσης θέσεων εργασίας, το οποίο όμως θα απαιτήσει μεγαλύτερη προσπάθεια ιδιαίτερα στην ε, ανισορροπία, αν θέλετε, δεξιοτήτων. Εγώ πιστεύω έντονα ότι δεν υπάρχει ε, πιο σοβαρή μορφή ε, ιεραρχίας διακρίσεων. Πιστεύω ότι υπάρχουν πολλαπλές διακρίσεις και πιστεύω ότι δεν υπάρχει ένα σαφές νομικό πλαίσιο, νομοθέτημα, διάταξη και λόγω του κατακαιρματισμού των κανόνων και των προτύπων στα κράτη-μέλη υπάρχει απόλυτη έλλειψη σαφήνειας. νομίζω επίσης ότι χρειαζόμαστε λίγο περισσότερο χρόνο για να εξετάσουμε όλες τις τροπολογίες που υπευλήθησαν. Έχουμε και 30 συμβαστικές από ό,τι κατάλαβα που είναι σημαντικός αριθμός. Είμαι υπέρ της αναβολής της συνάντησης των σκιωδών αλλά πρέπει επίσης να σας πω ότι εγώ δεν θα μπορέσω να έρθω την Πέμπτη γιατί έχω μια άλλη δέσμευση και θα ήθελα να ζητήσω να αναβληθεί πέραν της Πέμπτης για να μας δώσει και λίγο περισσότερο χρόνο για να μπορέσουμε να εξετάσουμε ενδελεχώς όλες τις συμβαστικέ, ώστε να έχουμε μια συνολική καλή εικόνα και κατανόηση της ε, γνωμοδότησης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Ο σκιώδης της Γκουέ. Έχουμε κάποιον. Δεν βλέπω. Πάμε στους πράσινους. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και την Ρενάτε Βέμπερ για μια πολύ καλή εγγνωμοδότηση και να πω δύο λόγια για τις τροπολογίες μας. Οι δικές μας όπως και της κυρία Στίβενς αφορούν εις τους ανθρώπους με αναπηρία το εκτιμώντα H, το 13α το 14 και οι προτάσεις για την νέα παράγραφο 13α είναι σύντομη και θα ήθελα να τη διαβάσω. Η αγορά εργασίας θα πρέπει να προσαρμόζεται περισσότερο, καλύτερα, στις ανάγκες των ανθρώπων με αναπηρία. Πρόκειται για μια στρατηγική, αν θέλετε, τοποθέτηση και προσέγγιση που θα θέλαμε να τονίσουμε μέσω της τροπολογίας αυτής. Επίσης, μια τροπολογία στην παράγραφο 14α σχετικά με την ενθάρρυνση προς τα κράτη-μέλη για την ενίσχυση των εργοδοτών που προσφέρουν θέσεις εργασίας σε ανθρώπου με αναπηρία. Χρειάζεται λοιπόν κατάλληλη υποστήριξη σε όλη τη διάρκεια της απασχόλησης. Και στο 15α σχετικά με την ε, αντιμετώπιση των διακρίσεων που υφίστανται οι άνθρωποι με αναπηρίες. Ε, μία άλλη δέσμη τροπολογιών αφορά εις τους ηλικιωμένους που δεν αναφέρονται πάντοτε στο πλαίσιο των διακρίσεων. Αλλά θεωρούμε ότι στο χώρο της εργασίας αυτό είναι σημαντικότατο πρόβλημα. γιατί οι ηλικιωμένοι δηλαδή λίγο πριν τη συντάξιμη ηλικία δυσκολεύονται ιδιαιτέρως να βρουν άλλη θέση απασχόλησης. Στην παράγραφο λοιπόν 19 πρέπει να τονίσουμε ότι χρειαζόμαστε αξιόπιστα στατιστικά δεδομένα σχετικά με τις δημογραφικές τάσεις και αλλαγές ώστε καλύτερα να έχουμε ε, ενεργείς ε, στρατηγικές ε, σχετικά τη, με την τρίτη ηλικία. Χρειαζόμαστε επίσης την πρόθεση του σχεδιασμού του περιβάλλοντος του εργασιακού που θα είναι πιο φιλικό για τους πιο ηλικιωμένους εργαζομένους. Επίσης υποβάλαμε μια τροπολογία σχετικά με τα στατιστικά δεδομένα gathering για την ανεργία, το οποίο θα έπρεπε να συζητηθεί. Αλλά λέμε ότι συλλέγοντας τέτοια δεδομένα προτείνουμε να συμπεριλαμβάνονται κάποιες προαιρετικές ερωτήσεις μιας διεργασιακής μελέτης για διακρίσεις επί τη βάση του φίλου της θρησκείας, της ιδεολογίας, της σεξουαλικής, του σεξουαλικού προσανατολισμού. που προκύπτουν από την οδηγία και από την χάρτα. Ε, με χαρά να, να συζητήσουμε το θέμα αυτό και με τους άλλους σκιώδεις Αυτές ήταν οι βασικές ιδέες από πλευράς μας. Thank you. I'll give... Ευχαριστώ. Σκιώδηση αυτή τη. Λαουράτζα. E ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και την Ρενάτε για την εξαιρετική της δουλειά από την αρχή εμείς έχουμε ασκήσει κριτική επί της ουσίας της οδηγίας. Η αντιμετώπιση των διακρίσεων εν πωλής είναι κάτι το σημαντικό, αλλά δεν πρέπει να αγνοούμε το βασικό κομμάτι των διακρίσεων που είναι οι διακρίσεις στο χώρο εργασίας. Αυτό είναι κάτι το οποίο μας κινητοποιεί, αν θέλετε, ιδιαίτερα. Εκφράζω λοιπόν την ευαρέσκειά μου γιατί η Ρενάτε προσπάθησε να συγκεντρώσει την προσοχή της ακριβώς στο χώρο εργασίας. Οι δικές μας τροπολογίες θέλουν να καλύψουν το θέμα αυτό. Η έκθεση της συναδέλφου Στίβενς ασχολείται με τα προβλήματα της αναπηρίας με ικανοποιητικό τρόπο και δεν ξέρω ε, αν θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο ίδιο επίπεδο και σε αυτήν την έκθεση. Εγώ θα ήθελα επίσης ε, να υπογραμμίσω ε, ένα επιπλέον θέμα το οποίο εμποδίζει τους ανάπηρους εργαζομένους πάρα πολύ συχνά ε, οι επιχειρήσεις προτιμούν να πληρώνουν τα πρόστιμα για τη μη πρόσληψη των αναπήρων παρά να προσαρμόσουν τις θέσεις εργασίας τους στους εργαζομένους με αναπηρίες. Είναι μία από τις χειρότερες διακρίσεις που μπορούμε να συναντήσουμε. Μέσω των τροπολογιών μας εμείς ε, είπαμε ότι υπάρχουν ε, τμήματα εργαζομένων που αποκλείονται από την αγορά εργασίας γιατί ούτε είναι σε συνταξιοδοτική ηλικία, ούτε είναι και νέοι, δηλαδή οι άνθρωποι γύρω στα 60 είναι αυτοί που βρίσκονται ένα βήμα πριν την έξοδο και για αυτούς θα πρέπει να προβλεφθούν δυνητικά συνοδευτικά μέτρα έτσι ώστε να μπορέσουν να εργαστούν εκ νέου. Έχουμε όλο και περισσότερους εργαζομένους οι οποίοι παραμένουν στις θέσεις εργασίας τους γιατί η κανόνες συνταξιοδότησης σκληραίνουν και αυτό δημιουργεί ε, μια προβληματική θα έλεγα η οποία δεν μπορεί να αγνοηθεί. Υπάρχουν ε, λοιπόν πολλές μορφές διακρίσεων οι οποίες θα πρέπει να συζητηθούν. Αγγλικά λέει η ομιλήτρια το stalking και το mobbing, δηλαδή η παρενόχληση, ο εκφοβισμός, η αδυναμία προστασίας αυτών που κάνουν καταγγελίες για το κοινό καλό. Νομίζω ότι απαιτούνται πολλές αλλαγές σε πολιτισμικό επίπεδο στην Ευρώπη και θα πρέπει με τις αλλαγές αυτές να προστατεύσουμε και τους καταγγέλλοντες. Ξέρετε ότι έχουν ξεκινήσει δικαστικές διαδικασίες σε πάρα πολλές χώρες μέλη για τέτοια προβλήματα οι διαδικασίες αυτές κρατούν ολόκληρα χρόνια, ενώ θα έπρεπε να ζητήσουμε οι διοικητικές διαδικασίες σχετικά με τις διακρίσεις να επιταχυνθούν και από την άλλη να προστατεύουν ε, τα συμφέροντα των εργαζομένων. Πάρα πολύ συχνά οι εργαζόμενοι δεν κάνουν βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση διότι δεν προστατεύονται δεν προστατεύονται τα προσωπικά τους δεδομένα, δεν προστατεύεται ο εμπιστευτικός χαρακτήρας των στοιχείων της κατάστασής τους. Στη δική μου χώρα το πρόβλημα αυτό υπάρχει. Υπάρχει νόμος, ο οποίος λέγει ότι για τους αναπήρους σαν παράδειγμα πρέπει να ξεπεραστούν τα εμπόδια που υπάρχουν και οι τροχοπέδες που υπάρχουν στην πλήρη άσκηση των δικαιωμάτων των ανθρώπων με αναπηρίες κτλ. Νομίζω ότι οι προσπάθειες πάντως της Ρενάτε είναι θετικές. Την ευχαριστώ γι' αυτό και ελπίζω να προχωρήσουμε σωστά. Σας ευχαριστώ. Μπιζότο δεν είναι εδώ η κυρία Μπιζότο, ο κύριος Μαρτά είναι εδώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Και συγχαρητήρια κυρία Βαμπέρη για την έκθεση. Δεν έχουμε καταθέσει τροπολογίες. Βεβαίω θα παρακολουθήσουμε και θα μελετήσουμε προσοχή ό,τι προτείνεται. Και γιατί γιατί η καταπολέμηση των διακρίσεων στην ε, εργασία, στην απασχόληση λόγω αναπηρίας, φίλου, θρησκείας, ηλικίας, βεβαίως και πρέπει να προχωρήσει. Στην αναπηρία είναι βεβαίως αυτονόητο ότι θα, θα βοηθήσουμε, θα στηρίξουμε κοινωνικά και θα, θα βοηθήσουμε στην ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας των, ε, το άτομο με αναπηρία αλλά όπως υπόθηκε και τώρα, ένα, μια κυρωτική προσέγγιση, τιμωρητική προσέγγιση έχει επιλεγεί. Εάν δηλαδή δεν προσλαμβάνει άτομο με αναπηρία μια επιχείρηση, θα έχει κυρώσεις. Καθώς όμως ε, πιστεύουμε είναι καλύτερη η ανταμοιβή, αφού τελευταία ανάλυση ο είναι εκείνος ο οποίος θα αποφασίζει, μια ανταμοιβή, ίσως φερειπίν με φοροαπαλλαγή, θα του φανεί ενδιαφέρουσα και θα τον οδηγήσει στην πρόσληψη ατόμων με αναπηρία για την ηλικία. Ό,τι και να λέτε. Πάλι ο εργοδότης είναι αυτός, ο διευθυντής μιας επιχείρησης είναι αυτός ο οποίος θα αποφασίσει και ό,τι και να λέμε ο νέος εργαζόμενος και λιγότερα θα του κοστίσει και καλύτερε επιδόσεις θα έχει και θα είναι πιο ικανός στη δουλειά του λόγω των ψηφιακών δεξιοτήτων. Αντίστροφα για τον ηλικιωμένο. Πρέπει λοιπόν και εμείς να αντιστρέψουμε το πρόβλημα και να αντλήσουμε τα ωφέλη της εμπειρίας των ε, πιο ηλικιωμένων μας, της τεχνογνωσίας δηλαδή που αποτελεί χρήσο ρηχείο, πλούτο τεράστιο. Και γι' αυτό νομίζω Πρέπει να ενθαρρύνουμε τους εργοδότες να κρατήσουν τους πιο ηλικιωμένους εργαζομένους για να μπορέσουν αυτοί να μεταγγίσουν, να μεταδώσουν τη τεχνογνωσία τους. Πάλι με ευεργετήματα κοινωνικά ή φορολογικά. Και βέβαια με την ιδέα ότι ο ηλικιωμένος θα πάρει υπό την ε, ε, αιγίδα του, υπό την προστασία του τον νέο εργαζόμενο. Έτσι θα κερδίσει και ο εργοδότης και οι εργαζόμενοι αλλά και τα ασφαλιστικά ταμεία, κυρίως τα ταμεία ανεργίας Σε σχέση με το φύλλο και την, ε, το χρόνο της ανεργίας, που είναι πολύ πιο περίπλοκα ζητήματα, βεβαίως δεν πρέπει να υπάρχουν διακρίσεις ε, στην ε, θρησκεία, επιστρέφω. Δεν πρέπει να υπάρχουν διακρίσει ούτε για τη λόγω θρησκεία ούτε λόγω σεξουαλική προτίμηση. Δεν πρέπει όμω και να πέσουμε σε ένα σύστημα θετικών προτιμήσεων. ει βάρο άλλων κοινοτήτων, να το πω έτσι. Εμεί θεωρούμε ότι κάθε αναγνωρίσιμη κοινότητα είναι η εθνική κοινότητα. η σεξουαλική, ο σεξουαλικός προσανατολισμό και οι θρησκευτικέ προτιμήσεις, επιλογές ανήκουν στην ιδιωτική σφαίρα και δεν μπορούν να οδηγήσουν σε καμία διάκριση. Και καταγγέλουμε σε αυτό τις θετικέ προτιμήσει που βλέπουμε και με την εκδήλωση του δικαιώματο τη ψήφου και με τις αλλαγέ σε να ε, να οδηγούν σε έκφραση αντιδράσεων, γιατί αυτοί οι οποίοι υπήρχαν τι συνέπειε αυτών των προτιμήσεων αντιδρούν όλο και περισσότερο και οργίζονται με τις κυβερνήσεις του και αυτό θα καθίσταται όλο και πιο εμφανέ. Είναι πολύ επικίνδυνα όλα αυτά που γίνονται, φερειπήρια ενσωμάτωση των πολιτικών προσφύγων με όρους πολιτικών ε, ε, προτιμήσεων στην αγορά εργασίας. Thank you, Mr. Koch. Ευχαριστώ, Κοχ. Είχατε το λόγο. Κυρία Βέμπερ, ήθελα καταρχάς να σε ευχαριστήσω για την πολύ καλή σας ε, έκθεση, το σχέδιο εκθέσεως. Η οδηγία για την ποιότητα στην απασχόληση είναι πολύ σημαντικό θέμα και σε αυτό θα πρέπει να συνεχίσουμε τη δουλειά. 18 ήταν δικές μου τροπολογίες από τις 314. Σημαντικές από αυτές είναι καταρχάς ότι το Κοινοβούλιο πάντοτε αγωνιζόταν κατά της εισαγωγής μιας ε, εγκάρσιας οδηγίας που θα απαγόρευε συλλήβδην της ε, διακρίσης γιατί θεωρεί ότι δεν θα ήταν δυνατό να υλοποιηθεί κάτι τέτοιο. Άρα θα πρέπει να εισάγεται η έννοια τη απαγόρευσης των διακρίσεων σε κάθε νομοθέτημα σχετικό με την εργασία. Επίσης θα πρέπει να εξασφαλίζεται ένα πεδίο ε, εργασίας κατάλληλο, ε, όχι με γενικούς όρους όμως, γιατί οι γενικοί όροι είναι ελάχιστοι όροι και ισχύουν και για τα άτομα με αναπηρία. Τα άτομα με αναπηρία όμως έχουν ειδικέ ανάγκες και ως εκ τούτου χρειάζονται ειδικό περιβάλλον. Ατομικά προσδορισμένο με βάση ατομικές τους ανάγκες περιβάλλον εργασίας. Μόνο έτσι μπορούν να έχουν ισότιμες ευκαιρίες εργασίας. Τρίτον, δεν θα πρέπει να ε, ζητούμε στατιστικές για ισότιμη μεταχείριση, αλλά αντικειμενικά αξιόπιστα δεδομένα για άνηση μεταχείριση, περιπτώσεις διακρίσεων και έτσι θα έχουμε και λιγότερη γραφειοκρατία. Επίσης, θα πρέπει και το κράτος να στηρίζει τα ε, ε, θύματα των ε, διακρίσεων βεβαίως, αλλά νομίζω ότι είναι υπερβολικό να μιλούμε για απαλλαγή από φόρο για τα θύματα των διακρίσεων και γι' αυτό ζητώ σχετική αναφορά να διαγραφεί. Κατά τα άλλα, ευχαριστώ και εύχομαι κάθε επιτυχία στη δουλειά σας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κώσα έχει το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο ήθελα καταρχάς να απευθύνω συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Στο παρελθόν είχαμε αρκετές φορές την ευκαιρία να συνεργαστούμε στα θέματα αυτά. Έχω την εμπειρία λοιπόν και την οσιοδοξία ότι θα έχουμε πολύ καλές συμβαστικές λύσεις και σε αυτή την ε, οδηγία, σε αυτήν την έκθεση. Έχουμε να κάνουμε με μία προσέγγιση της ε, καταπολέμησης των διακρίσεων σε σχέση με τα άτομα με αναπηρία και δεν νομίζω ότι τα άτομα με αναπηρία θα πρέπει να είναι αυτά που θα πρέπει να φέρουν το βάρος της διάκρισης. Είναι κοινή η ευθύνη, κοινό το βάρος. Πιστεύω λοιπόν ότι δεν έχουν ε, προχωρήσει όλα τα κράτη όπως όφυλαν στην υλοποίηση της οδηγίας μέχρι τώρα Γι' αυτό και η δουλειά του Κοινοβουλίου είναι πολύ σημαντική. 310 είπαμε είναι οι τροπολογίες. Αυτό δείχνει πόσο πολύ ενδιαφέρει το Κοινοβούλιο η υπόθεση αυτή και πόσο θέλει να καταστήσει πιο αποτελεσματική την εφαρμογή της οδηγίας. Όλοι οι προλαλήσαντες υπεγράμμισαν τη σημασία της καταπολέμησης των διακρίσεων εις βάρος ατόμων με αναπηρία. Εγώ ως άτομο με αναπηρία ο ίδιος θέλω να επισημάνω ότι δεν πρέπει να πάμε και πολύ μακριά. Βεβαίω έχει στρατευτεί υπέρ των ατομών με αναπηρία το Κοινοβούλιο, αλλά πρέπει να δείξει ότι χρειάζεται να καταπολεμηθούν οι διακρίσεις σε κάθε τομέα, είτε πρόκειται για θρησκεία, είτε πρόκειται για σεξουαλική προσανατολισμό, ηλικία, ε, αναπηρία και πολλούς άλλους τομείς στους οποίους πάλι πρέπει να επαγρυπνούμε κατά των διακρίσεων. Και εγώ Έχω καταθέσει πολλές τροπολογίες επιτοπλίστων κατά των διακρίσεων. Τροπολογίες όμως οι οποίες ε, κυρίως αφορούν άλλες κοινωνικές κατηγορίες και θα ήθελα να αναφερθώ στο ζήτημα της ε, ορθολογικής εμπλοκής ε, πρόκειται για την τροπολογία 208 και ελπίζω να την υποστηρίξει η συγγήτρια. Δηλαδή εδώ μιλάμε για μια προσαρμογή ορθολογική, 108 τροπολογία, επανέρχομαι. Και βέβαια μιλούμε για τα άτομα με αναπηρία, αλλά αφορά όλα τα θύματα ε, διακρίσεων και σημαίνει αυτό καλύτερες υπηρεσίες στο χώρο εργασία. Και ταυτόχρονα, και ενώ μπορεί να φαίνεται εκ πρώτης αφορά τα άτομα με αναπηρία, ε, οπωσδήποτε έχει να κάνει με οποιονδήποτε κατά τη διάρκεια του επαγγελματικού του βίου αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας, αρρώστια, είναι αυτό ή ατύχημα. Τι θέλω να πω συγκεκριμένα, ότι μόνο με ιατρικό πιστοποιητικό μπορεί κανείς να επικαλεστεί ασθένεια στις προσθέρες χώρες. Ευτυχώς η χώρα μου η Ουγγαρία δεν είναι ε, μια από αυτές βεβαίως και λαμβάνονται υπόψη το ιατρικό πιστοποιητικό, αλλά ταυτόχρονα εξετάζονται και ή δυνατότητες στην ουσία να εργαστεί ο ενδιαφερόμενος και με βάση τις δυνατότητες που έχει στην διάθεσή του και τις ικανότητες προς εργασία γίνεται η προσαρμογή στις εργασιακές συνθήκες. Αυτά λοιπόν και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να έχουμε έτσι μια βελτίωση της οδηγίας. Thank to Θέλετε να προσθέσετε κάτι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις που ζήτησαν το λόγο, να τους ευχαριστήσω για τα θετικά τους λόγια, αλλά να τους ευχαριστήσω επίσης και για την ουσιαστική συνεισφορά τους. Από αυτά τα οποία άκουσα μέχρι τώρα μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι πολλές από τις ιδέες αυτές έχουν ήδη ενταχθεί στις συμβιβαστικές τροπολογίες. Ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησαν οι συγκεκριμένες τροπολογίες, αλλά εγώ επέστρεψα μετά από μια αποστολή σχεδόν τριών εβδομάδων στο Περού. Ήταν λοιπόν πάρα πολύ δύσκολο να έχω επικοινωνία μαζί σας πέραν του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Γι' αυτό λοιπόν λάβατε τις, θα λάβετε μάλλον τις συμβιβαστικές στις 12 το μεσημέρι. Πέρα από την διαδικασία Νομίζω ότι μία από τις προτάσεις θα ήταν να υπάρξει μια συνάντηση πράγματι την Πέμπτη για να συζητηθεί ο μισός αριθμός των τροπολογιών και την επόμενη εβδομάδα για τις υπόλοιπες. Εγώ είμαι εδώ και την εβδομάδα αυτή και την επόμενη εβδομάδα θα είμαι συνεχώς εδώ ε, και την μεθεπόμενη νομίζω ότι έχει σημασία να καταλήξουμε σε κάποιες από τις συμβιβαστικές τις οποίες θα σας καταθέσω. Τώρα, επί της ουσίας επαναλαμβάνω, πολλά από αυτά τα οποία είπατε είναι πράγματα τα οποία κάλλιστα θα μπορούσα να δεχτώ. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει ιεραρχία σε σχέση με τις διακρίσεις και ότι τα πιο επικίνδυνα πράγματα Unfortunately, is a daily reality. Ε, το θέμα είναι ότι η πραγματικότητα μας ε, δεν μας διαψεύδει, μας επιβεβαιώνει καθημερινά. Μία από τις βασικές ιδέες είναι ότι um, uh, uh, Υπάρχει το θέμα της καταπολέμησης ε, γενικά των διακρίσεων στο εσωτερικό της, του χώρου εργασίας. Δεν είναι μόνο αυτό όμως. Εάν πράγματι επιθυμούμε να μειώσουμε το επίπεδο των διακρίσεων και μάλιστα να απαλλαγούμε από τις διακρίσεις, θα πρέπει να υπάρξει μια ευρύτερη αντιμετώπιση, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις διακρίσεις σε όλους τους τομείς, όπως την εκπαίδευση. Και γι' αυτό η ιδέα μιας οριζόντιας οδηγίας είναι μια νομίζω καλή ιδέα και έχει εκφραστεί από πάρα πολλούς ε, από όσους πήραν το λόγο μέχρι τώρα. Λοιπόν, ελπίζω οι συζητήσεις που θα ακολουθήσουν να είναι καρποφόρες και να καταλήξουμε σύντομα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. 21 Απριλίου στην Επιτροπή και ελπίζω να φτάσουμε στο Ολομέλεια τον μήνα Σεπτέμβριο μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Σας ευχαριστώ. Συνεχίζουμε με το σημείο 10 δημοσιονομικός έλεγχος της χρηματοδότησης των ΜΚΟ. Η κυρία το... έχει το λόγο. Το λόγο έχει η κυρία... Η κυρία Σδανόκα, η συγγετρία. Ευχαριστώ πρόεδρε. Να ευχαριστήσω... Employment για την ε, προπαρασκευαστική εργασία που έγινε όπου συνεργαστήκαμε με τη ΣΜΚΑ Όμικρον είχαμε μια σειρά από συναντήσεις και διαβούλευση με πολλές οργανές, οργανώσεις και με δίκτυα οργανώσεων και αποτυπώνεται αυτό στην πρότασή μας. Ε, λόγος εξάλλου για τον οποίο είναι και πολύ μεγάλη σημασίας, κρίσιμη σημασίας αυτή η γνωμοδότηση σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Κοινωνικής ε, Απασχόλησης και Καινοτομίας Βεβαίως οι περιορισμοί της έκθεσης δεν μας επέτρεψαν να καλύψουμε όλες απολύτως τις πτυχές του θέματος. Είχαμε βεβαίως προτάσεις και ελπίζω ότι όταν θα συνεργαστούμε με τους Κιώδης θα μπορέσουμε να καλύψουμε όλες τις ανησυχίες που ακούστηκαν από τους μη ΚΟ, με τους οποίους θα έρθουμε σε επαφή ώστε οι συστάσεις μας να είναι όσο το δυνατόν πλησιέστερες στις ανάγκες τους. Για τις ευρωπαϊκές κοινωνικές ΜΚΟ υπάρχει μια κάποια ευρωπαϊκή χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία υπάρχει όμως μια συνολική μείωση της χρηματοδότησης το οποίο μας οδηγεί στην πιο αποτελεσματική χρήση των υφισταμένων κονδυλίων. Και εδώ αντιμετωπίζονται δυσκολίες στην πρόσβαση προς τη χρηματοδότηση, όπως και στις απαιτήσεις, στις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων, τις διαδικασίες δηλαδή βάσει των οποίων λαμβάνει κανείς χρηματοδότηση. Επίσης υπάρχουν επιχειρησιακές χορηγίες που είναι κατά μέγιστον ενός έτους και για να πάνε πέραν του έτους χρειάζεται ενδείξεις ε, ε, συνέχειας του προγράμματος και βιωσιμότητας του προγράμματος. το οποίο σε κάποιες περιπτώσεις απειλεί το έργο των οργανώσεων αυτών ακριβώς τη στιγμή που είναι πιο απαραίτητο βάσει των συνθήκων που επικρατούν σήμερα. Υπάρχουν ομάδες πληθυσμού των οποίων τις ανάγκες μπορούν να βοηθήσουν και να καλύψουν μόνο τέτοιου είδους οργανώσεις. Και άρα πρέπει να πασχίσουμε για να εξασφαλίσουμε τη χρηματοδότησή τους. Μέσω του Ταμείου αυτού απασχόλησης κοινωνικής καινοτομίας. Ε, Μόνο δημόσιοι οργανισμοί, δημόσιοι φορείς μπορούν να υποβάλουν την πρότασή τους για να λάβουν χρηματοδότηση. Εμείς λοιπόν υποβάλλουμε μια πρόταση ώστε να τροποποιηθεί ο κανόνας αυτός και να μπορούν να ηγούνται των προγραμμάτων όχι μόνο δημόσιοι φορείς αλλά και μη καπαόμικρον. Σημειώνουμε επίσης ότι τα κονδύλια αυτά απαιτούν, προϋποθέτουν συγχρηματοδότηση. Και ένα πολύ υψηλό ποσοστό μπορεί να μην είναι εποφέλες για, τους, για τις οργανώσεις εκείνες που δεν θα μπορούσαν να φτάσουν σε ένα τέτοιο επίπεδο. Επίσης, το πεδίο αυτό καλύπτεται από διάφορες γενικές διευθύνσεις της Κομισιόν και καλούμε την Κομισιόν να συνδυάσει περισσότερα επιχειρησιακά κονδύλια από περισσότερες δηλαδή γενικές διευθύνσεις Αυτές είναι οι προτάσεις μας και με χαρά να ακούσω τις ιδέες και τις προτάσεις των σκιωδών για να ενσωματώσουμε τις προτάσεις αυτές ή στην γνωμοδότηση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ρωμανία Τόμ ε, από το ΕΛΚ. Ε, ευχαριστώ Πρόεδρε. <clears throat> Να ευχαριστήσω και εγώ την εισηγήτρια για τη δουλειά της. Στην γνωμοδότηση αυτή. Πιστεύω ότι έχουμε να κάνουμε με μια καλή, με ένα καλό σχέδιο γνωμοδότηση, μια καλή βάση εργασίας και πιστεύω όλοι συμφωνούμε πως οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην καθημερινή μας ζωή. Και ένα πολύ σημαντικό θέμα βέβαια είναι στη δουλειά των μη κυβερνητικών οργανώσεων η εθελοντική εργασία και οι εθελοντές. Οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς ε, των κοινωνιών μας. Είναι πολύ σημαντικό οι παράγοντες σε κάθε τομέα της ζωής είναι οι ίδιοι οι άνθρωποι, εκπροσωπούν τους πολίτες και ως εκ τούτου θα πρέπει να τις υποστηρίζουμε και οικονομικά και να ενθαρρύνουμε τη δουλειά τους. Όταν συζητούμε τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις, βεβαίως θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και την άλλη όψη, την άλλη εκδοχή δεν πρέπει να μιλούμε δηλαδή μόνο για δικαιώματα και θετικά στοιχεία ε, της δουλειά τους. Θα πρέπει να μιλούμε για τη δουλειά αυτή, η οποία πρέπει να είναι ισορροπημένη και όχι πολιτικοποιημένη ή κομματικοποιημένη, γιατί αυτό έχω δει στη Σλοβενία, την πατρίδα μου, ότι μερικές φορές αναλαμβάνουν δρόμο, ε, ρόλο πολιτικών ε, φορέων με κυβερνητικέ οργανώσεις και παίρνουν συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές, έστω και αν δεν το ομολογούν ανοιχτά. Και άρα δεν συμπεριφέρονται ως πολιτικά κόμματα, ενώ έχουν κάνει κομματικές επιλογές. Αυτό πρέπει να το υπογραμμίσουμε λοιπόν. Γιατί αν σημαίνει αυτό πρέπει να φέρουν και την ευθύνη της αντικειμενικότητας σε μη κυβερνητικές οργανώσεις. Έχω λοιπόν τα εξή ερωτήματα προς την εισηγήτρια. Πρώτον, πώς μπορούμε όλοι μας να συμβάλλουμε ώστε να εξασφαλιστεί η ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα των μη κυβερνητικών οργανώσεων, ιδιαίτερα όσον αφορά τα κοινωνικά. Ξέρω ότι βεβαίω είναι αδύνατο να εξασφαλιστεί σε απόλυτο βαθμό αυτό, αλλά θα πρέπει να προσπαθήσουμε και έχουμε δει κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα μη κυβερνητικών οργανώσεων που αξιοποιούν ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για να πολεμήσουν κάποια εγχειρήματα και έργα που πάλι έχει χρηματοδοτήσει ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός. Εδώ έχουμε να κάνουμε με μία ε, σύγκρουση συμφερόντων που θα πρέπει να εξουδετερωθεί. Και για να ολοκληρώνω. Θα ήθελα για άλλη μια φορά να πω ότι το σχέδιο γνωμοδότης αποτελεί πολύ καλή βάση για τη δουλειά μας. Βεβαίως θα εισαγάγουμε προτάσεις τροπολογίας εκ μέρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, αλλά βεβαίως θα μπορέσουμε να βρούμε και κάποιο κοινό πεδίο συνεννόηση. Ευχαριστώ της Δημοκράτες, κυρία Καηλίος Σκιώδης. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ Τατιάννα για την πολύ καλή δουλειά που έκανε στη συγγνωμοδότηση αυτή, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου έχει πολύ μεγάλη σημασία και έχει μεγάλη προβολή στα πρωτοσέλιδα όλες της Ευρώπης το θέμα της σωστής χρηματοδότησης των σωστών μη κυβερνητικών οργανώσεων και βεβαίως θα πρέπει να δούμε την, ε, τις συνέπειες ε, σε σχέση με τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Το Ταμείο για την υποστήριξη των πιο φτωχών δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς τη συμβολή των μη κυβερνητικών οργανώσεων και αυτές με την πλευρά τους δεν μπορούν να προσφέρουν έργο χωρίς να έχουν πόρους σε υλικό και ανθρώπινο κεφάλαιο. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει οι μη κυβερνητικέ οργανώσει να παίρνουν πάντα χρηματοδότηση και μόνο από τι κυβερνήσει. Πρέπει και αυτό να μα απασχολήσει στην έκθεση, που θα είναι δηλαδή το σημείο ισορροπία. Τρία στοιχεία θέλουμε να υπογραμμίσουμε. Πρώτον, ανάγκη όσο το δυνατόν περισσότερο να επιταχυνθεί η κοινωνική ε, ενσωμάτωση, εμπλοκή μάλλον των μη κυβερνητικών οργανώσεων σε καταστάσεις ε, βεβαίως πάγιες αλλά και σε επίγουσες καταστάσεις για να βελτιστοποιηθεί αυτή η εμπλοκή θα πρέπει να δημιουργηθεί, γιατί δεν υπάρχει ένας απλός διαφανής ε, μηχανισμός, ένα πλαίσιο το οποίο θα επιτρέπει με απλούς τρόπους την ανταπόκριση σε προβλήματα κατεπήγοντα όπως αυτά τα οποία αντιμετωπίζει η Ευρώπη στα νοτιοανατολικά της, Επίσης θα πρέπει να έχουμε ευέλικτη και υπεύθυνη ανταπόκριση στις ανάγκες των κυβερνητικών οργανώσεων ώστε όταν υπάρχουν ανάγκες απρόβλεπτες να μπορούν να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά. Είναι απαραίτητο βεβαίως να υπάρξει κατάλληλη χρηματοδότηση για να εξασφαλίζεται το απαραίτητο κεφάλαιο και μέσα για τους παράγοντες αυτών των κυβερνητικών οργανώσεων που μπορούν να δράσουν επικοδομητικά σε, μέσο και μακρο, σε βράχη και μέσο πρόθεσμο ορίζοντα, κυρίω για του ανθρώπου των οποίων ζωτικέ ανάγκε χρειάζονται κάλυψη και βεβαίω θα θέλαμε με τη γνωμοδότηση να καλυφθεί και η ανάγκη για διαλειτουργική σχέση μεταξύ των προγραμμάτων χρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και εκείνων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, δεδομένου ότι Πολύ συχνά οι μη κυβερνητικέ οργανώσει ε, απασχολούνται από τι κυβερνήσει, όχι απαραίτητα πάντα με διαφανεί διαδικασίε, παραμένουν εκτό υποχρέωση λογοδοσία και εκτό ελέγχου, ανεξαρτήτω του αν υλοποιούν ε, τα υπεσχημένα. Και έτσι το να χορηγούνται, για να χορηγούνται οι πόροι κατά τρόπο εύθετο, έγκαιρο και αντικειμενικό, σημαίνει και εξασφάλιση των μέγιστων αποτελεσμάτων, αξιοπιστίας και όφελος μόνο προς τις ε, σωστές και αψεγάδια στις μη οργανώσεις και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα και όχι απλώς περιγραφές στόχων ή κάποια δοκίμια που μπορεί να παρουσιάσουν έκθεση, μια έκθεση ιδεών, αλλά με πραγματικά αποτελέσματα, γιατί πολλές φορές βλέπουμε μη κυβερνητικέ οργανώσεις να αυτοανακηρύσσονται εθελοντικές, ενώ έχουν έντονο συσχετισμό με τις τοπικές μαφίες και τη διευκίνηση ακόμη ανθρώπων, όπως ε, την Κυριακή ε, είδαμε αυτή την Κυριακή στις ειδήσει στην Ελλάδα σε σχέση με την προσφυγική κρίση ότι υπάρχουν μη κυβερνητικέ οργανώσεις οι οποίες αξιοποιούν χρηματοδότηση ενώ βρίσκονται ακόμη υπό διερεύνηση αστυνομική ακόμη και για απάτη και εξακολουθούν να σπράττουν τη χρηματοδότηση και είναι εμπλεγμένε με μαφίε που διακινούν ε, πρόσφυγες, αλλά πάλι εξακολουθούν να εισπράττουν χρηματοδότηση από κυβερνήσεις και ταυτόχρονα ε, έχουν υπό τον πλήρη έλεγχό τους τις καταστάσεις, τις χειραγωγούν τις καταστάσεις αυτές και τις διαιωνίζουν με εντάσεις που προξενούν προκειμένου να εξακολουθούν να εισπράττουν χρηματοδότηση, δηλαδή να διατηρούν το λόγο ύπαρξής τους στην ε, περιοχή. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να δώσουμε απαντήσεις. Ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο το έργο σου. ευχαριστώ θερμά για τις προσπάθειές σου και η διαφάνεια πιστεύω πρέπει να είναι το σημείο εστιαση. Θα συνεχίσουμε βεβαίω και με τι τροπολογίε. Ευχαριστώ θερμά. Thank you. Mr. E Ευχαριστούμε. Ο εκπρόσωπος του ECR, η κυρία Ντρεσίνσκα δεν είναι εδώ. Όχι. Πάμε στην Άλντε. Η κυρία Χάρκιν, ευχαριστώ πρόεδρε και να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τη συνάδελφο για μια πολύ καλή βάση για την γνωμοδότηση για τις κοινωνικές ομικρον ε, Συμφωνώ με την εισηγήτρια ότι η κοινωνική αποστολή των οργανώσεων αυτών είναι ευάλωτη τώρα που έχει μειωθεί η χρηματοδότησή τους και είναι πολύ σημαντική η δουλειά τους και τη χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή. Σε προηγούμενες περιπτώσεις αυτές ε, οι υπηρεσίες καλύπτονταν από δημόσιες υπηρεσίες που αυτή τη στιγμή έχουν συρρυκνωθεί για διάφορους λόγους. Μαζί με τα σλοβενικά και ελληνικά σχόλια θα ήθελα να προσθέσω και μερικά από πλευράς μας Ιρλανδικά ε, σχετικά με κάποιες καταστάσεις που ενδεχομένως να μην γνωρίζουμε αλλά είναι καλό να έχουμε μια συνολική εικόνα για το τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Οι περικοπές στη δική μας χώρα έχουν οπωσδήποτε επιφέρει αντίκτυπο σε πάρα πολλές κοινωνικές μικρών και την ικανότητά τους να καλύπτουν τα πεδία ιδιαίτερα της ε, κοινωνικής ε, ένταξης που είναι πολύ σημαντική. Χρειάζεται λοιπόν να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη για να βοηθήσουν τις καπα-όμικρον σε συγκεκριμένα πεδία πολιτικής. Ε, δεν έχω καμία αφιβολία ότι αυτό διαφέρει πολύ από χώρα σε χώρα, αλλά πολύ συχνά έχουμε την ψευδέστηση ότι έχουμε επιτύχει μια κοινωνική συνοχή και ενσωμάτωση. Είμαι απολύτως υπέρ ε, της ε, διατύπωσης στην παράγραφο 3 σχετικά με την ανεξαρτησία των ΜΚΟ και ίσως εκεί να έχουμε διαφορετικές ε, προσεγγίσεις. Ε, θεωρώ όμως ότι ο ρόλος που δεδοματίζουν οι ε, είναι κρίσιμος. Πρέπει να είναι ναι αντικειμενικές, αλλά όχι σιωπηλέ. Έχουν πολλή δουλειά να κάνουν στη συλλογή πληροφοριών, σε διάφορες εξτρατείες ευαισθητοποίησης και ίσως στη συμμετοχή τους στην πολιτική σκηνή, αλλά με μικρό και όχι κεφαλαίο όπως θα το έλεγα. Είμαι από εκείνους που είναι απολύτως υπέρ της συμμετοχικής δημοκρατίας και σε αυτό το πεδίο η καπαόμικρον διαδραματίζουν σημαντικότατο ρόλο. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε εδώ να βρούμε μια διατύπωση που θα είναι αποδεκτή από όλους. Μίλησε η συγγήτρια για την δυσκολία που αντιμετωπίζουν στην χρηματοδότηση, στην πρόσβαση στη χρηματοδότηση, τις προϋποθέσεις και τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων κτλ διότι πάντοτε μεταξύ της πλευράς του ελέγχου και της επιχειρησιακής πλευράς ε, χρειάζεται μια ισορροπία. Και πολύ συχνά ακούμε παράπονα και από μη καπαόμικρον και από άλλους φορείς σχετικά με την περιπλοκότητα των διαδικασιών υποβολής και κάθε φορά πρέπει να πατήσουμε το πράσινο ή το κόκκινο ή το λευκό κουμπί για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Αυτό είναι μια δική μας ευθύνη. Και θα πρέπει να βρούμε έναν σωστό και καλό τρόπο. Ακούσαμε και τα σχόλια από την Ελληνίδα συνάδελφο για το πώς μπορούν να αποκλίνουν τα πράγματα. Δεν πρέπει να προσθέτουμε στην περιπλοκότητα. Πρέπει να το προσέχουμε όσο μπορούμε αυτό το σημείο. Είμαι βέβαιη ότι μπορούν να γίνουν βελτιώσεις. Συμφωνώ επίσης σχετικά με το γεγονός ότι πρέπει να πάμε πέρα από το σύστημα χορηγίας μονοετούς και να δούμε κάποια πολυετή προγράμματα τα οποία απαιτούνται για να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα της δραστηριότητας. Και συμφωνώ με την συνάδελφο που αναφέρθηκε στον εθελοντισμό και πόσο σημαντική είναι αυτή η δουλειά. Επιφέρει τεράστια προσταθέμενη αξία. Πάρα πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά χωρίς την συμμετοχή των εθελοντών. Και για να κλείσω, όπως ξεκίνησα, άκουσα τους συναδέλφους ε, από την ομάδα των σοσιαλιστών και το ΕΛΚ ε, σχετικά με τις καταχρήσεις και την εκπετάλευση που πολλοί φορείς επιχειρούν να επιφέρουν ή να χρησιμοποιήσουν εγώ ακούω τους συναδέλφους, ελπίζω ότι θα μπορέσουμε όμως να βρούμε μια διατύπωση ε, που θα ικανοποιεί άπαντης. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω για την γνωμοδότηση. Καλύπτει πολλές από τις ανησυχίες τις οποίες είχαμε. Θα συμφωνήσω επίσης ότι η προκυκλική φύση των δαπανών αυτών σε σχέση με την χρηματοδότηση των δαπανών τους οδηγεί σε περικοπές και μάλιστα μια εποχή όπου οι υπηρεσίες τους είναι ιδιαίτερα χρήσιμες. Θα πρέπει φυσικά οι ΜΚΟ να έχουν την δυνατότητα να εκφράζονται ελεύθερα έχουν πάρα πολλά προβλήματα επιμελητιακά να αντιμετωπίσουν, είναι στα πλαίσια των ευθυνών τους αυτό. Τα προγράμματα χρηματοδότησης είναι ιδιαιτέρως περίπλοκα, γραφειοκρατικά και χρονοβόρα. Και αυτό είναι ένα βασικό πρόβλημα για πάρα πολλές ΜΚΟ με τις οποίες έχω συναντηθεί. Θα πρέπει εδώ να υπάρξει ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να υπάρξει μια αντιμετώπιση των προβλημάτων εκ των κάτω προς τα πάνω, έτσι ώστε να υπάρχει σωστή αντίληψη για τα προβλήματα και επίσης θα πρέπει να υπάρξει και χρηματοδότηση αν είναι δυνατόν σε πολυετή βάση και όχι σε αυστηρά ετήσια. Υπάρχει παράλληλα και το θέμα της συγχρηματοδότησης. Ένα από τα προβλήματα που εμείς αντιμετωπίζουμε στη δική μου χώρα, στην Ιρλανδία, είναι οι αλλαγές πηγών χρηματοδότησης και εδώ το θέμα της αντιμετώπισης του προβλήματος εκ των κάτω προς τα πάνω θα μπορούσε να προσφέρει λύσεις. Προσπαθούμε ε, με τις τροπολογίες μας να υπογραμμίσουμε τα σημεία τα οποία περιλαμβάνει έτσι και αλλιώς η γνωμοδότηση, ιδιαίτερα για την ανάγκη της ανάπτυξης ε, του τρόπου χρηματοδότησης των ΜΚΟ. Οι ΜΚΟ έχουν, ε, έχουν την δυνατότητα να επηρεάσουν σε κοινωνικό επίπεδο την κατάσταση μακροπρόθεσμα, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο να φανεί και να αντικατοπτριστεί σωστά σε αιτήσια βάση, σε επίπεδο ισολογισμού ή απολογισμού των δραστηριοτήτων τους. Συνεπώς θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε, έστω και με δύσκολο τρόπο, πόσο ποιοτικά επηρεάζουν και αποδίδουν οι συγκεκριμένες ΜΚΟ. Ευχαριστώ κυρία Τζία. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την Τατιάνα για την πολύ καλή δουλειά της. Την ευχαριστούμε γι' αυτό και θα συνεργαστούμε με χαρά μαζί της. Συμφωνώ με το τελευταίο σημείο, ο, προκυκλικός χαρακτήρας η πορεία του ΑΕΠ της κάθε χώρας και οι δημόσιες δαπάνες ε, ε, εξαρτώνται πολύ από τις χρηματοδοτικές ικανότητες ε, των χωρών και επηρεάζονται οι ΜΚΟ. Έχω κάποια θέματα με το άρθρο 2 και με την λειτουργία των διαφροτικών και του κοινωνικού ταμείου και στο βαθμό που επιτρέπει την χρηματοδότηση των ΜΚΙΟ. Θα ήθελα να καταλάβω όταν λέτε ότι δεν μπορούν να υπάρξουν αλλαγές χωρίς την, να εφαρμοστούν μάλλον χωρίς την συμμετοχή των ΜΚΙΟ, αν αυτό είναι κάτι το οποίο εξαρτάται από τα προβλήματα που έχουν οι ίδιες οι ΜΚΙΟ να χρησιμοποιήσουν και διαφορετικές μορφές χρηματοδότησης. Θυμίζω το πρόγραμμα Progress για τις μικροπιστώσεις είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ε, θα έλεγα ε, θα μπορούσε να λειτουργήσει με πολύ χρήσιμο τρόπο και θα ήθελα να μου δώσετε εδώ κάποιες διευκρινήσεις. Θα συμφωνήσω επίσης ε, και για την ανεξαρτησία η οποία θα πρέπει να χαρακτηρίζει τις ΜΚΟ. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα έλεγα είναι εγγύηση για την αποστολή των ΜΚΟ και για την εκπλήρωση των στόχων τους και των εντολών τις οποίες έχουν. Όταν μιλάμε για μικιό να μην ξεχνάμε ότι θα πρέπει να μην ξεχνάμε και τις πολύ μικρές μικιό οι οποίες καταφέρνουν με συγκεκριμένο τρόπο να χρηματοδοτηθούν είναι οι μεγάλες μικιό. Οι μικρές όμως, οι ενώσεις, οι τοπικοί σύλλογοι που σε τοπικό επίπεδο κάνουν μια εξαιρετική δουλειά θα έπρεπε και αυτές να υπάρχει δυνατότητα να βοηθηθούν και να υποστηριχθούν. Ίσως να είναι χρήσιμο εδώ και η δημιουργία ενός database, μιας βάσης δεδομένων, ενός database των ΜΚΟ έτσι ώστε το θέμα της καταγραφής τους, ε, κάτι το οποίο είναι πρόβλημα, είναι περίπλοκη επίσης η συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς και προμήθειες δημόσιες. Πρέπει να βρεθούν τρόποι να υποστηριχθούν οι ΜΚΟ. Θα ήθελα επίσης να κάνω και ορισμένες παρατηρήσεις για την δυνατότητα που θα πρέπει να έχουν οι ΜΚΟ να ηγούνται στην παρουσίαση ενός προγράμματος που χρήζει χρηματοδότησης. Το να έχει κανείς μια ηγετική θέση από τη μία προσδίδει προς τη θέμενη αξία στην ΜΚΙΟ και ταυτόχρονα πολύ συχνά οι εταιρικέ σχέσεις ναι μεν ξεκινούν καλά αλλά να βαγούν διότι πολλές φορές υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ τους έστω και στη μέση της διαδικασίας. Συνεπώς η ηγετική ομάδα έχει διπλές ευθύνες και περιπλέκεται ο ρόλος και η λειτουργία τους. Ίσως λοιπόν θα πρέπει να διευκρινιστεί καλύτερα η διαδικασία και να βρούμε μια σωστότερη αν θέλετε διατύπωση για το συγκεκριμένο πρόβλημα. Δεν ξέρω αν ξέρετε πώς λειτουργεί ακριβώς ο κανονισμός του Horizon 2020 το πρόγραμμα αυτό έχει δημιουργηθεί για να υποστηριχθούν τα πανεπιστήμια και η έρευνα, η πανεπιστημιακή. Και προβλέπεται πολλές φορές η χρηματοδότηση για συγκεκριμένα προγράμματα κατά 100%. Ίσως θα πρέπει και σε αυτό το πλαίσιο και σε αυτό το επίπεδο να δώσουμε τις εγγυήσει στις ΜΚΟ, οι οποίες θα έχουν την δυνατότητα χρήσης αυτών των πιστώσεων σύμφωνα πάντα με τον κανονισμό του Horizon, Horizon 2020 και να αποφύγουν τα συστήματα συγχρηματοδότησης τα οποία είναι πολύ περίπλοκα. Γιατί επαναλαμβάνω ότι η ΜΚΟ είναι μη ε, κερδοσκοπικές οργανώσεις, οπότε ε, για τις μεγάλες ΜΚΟ πολλές φορές η χρηματοδότηση μεταφράζεται ακόμα και με ε, παροχή εργασίας δυνατοτήτων ορών εργασίας και έτσι καλύπτουν το κόστος λειτουργίας τους. Αυτό όμω ισχύει μόνο για τις μεγάλες ΜΚΟ. Οι μικρές ΜΚΟ δεν μπορούν να διευκρινίσουν το κόστος αυτό και δεν μπορούν να το χαρακτηρίσουν σαν ένα τμήμα του συνολικού κόστους εργασίας τους. Και τώρα για το σημείο 10 θα ήθελα να μάθω τι ακριβώς εννοείται ε, για την δημοσίευση των αποτελεσμάτων. Όταν κάποιος προσπαθεί να πάρει μέρος σε μια δημόσια προμήθεια, σε ένα διαγωνισμό ε, και αυτό ε, θα έλεγα περιλαμβάνεται σε πίνακες οι οποίοι καταρτίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η δημοσιοποίηση αυτού του πίνακα σημαίνει ότι θα δημιουργηθεί μια νέα βάση δεδομένων, σημαίνει ότι θα υπάρξει μια θα έλεγα σωστή ενημέρωση για τις χρηστές πρακτικές. Η βαθμολόγηση αυτή θα είναι ουσιαστικά ένα μέτρο για την αξιολόγηση της λειτουργίας τους. Εγώ νομίζω ότι ο ρόλος τον οποίο έχουν να παίξουν οι ΜΚΟ είναι πάρα πολύ σημαντικός. Πρέπει όμως να δώσουμε την δυνατότητα και στις μικρές ΜΚΟ που εργάζονται σε συγκεκριμένα εδάφη. Ξέρετε ότι σε χώρες όπως η Ελλάδα σαν παράδειγμα η υποστήριξη που δίδεται στους πρόσφυγες εν πολλής καλύπτεται από τις ΜΚΟ και κυρίως από πολύ μικρές ΜΚΟ. Κάποιοι φοιτητές που οργανώνονται σε μικρές ομάδες και κάνουν πάρα πολλά ε, για τα προβλήματα των ε, προσφύγων. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να δώσουμε μια διάσταση πιο περιορισμένη και πιο προσαρμόσιμη έτσι ώστε όλες οι ΜΚΟ να μπορέσουν να βοηθηθούν και να χρηματοδοτηθούν. Thank you. Ε, Ευχαριστώ. Κυρία Μάρτα, να ο κύριος Φούντολης την εκπροσωπεί. Παρακαλώ. Στον έλεγχο του προπολογισμού σχετικά με τη χρηματοδότηση των μη κυβερνητικών οργανώσεων από τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα προσέθετα και τον έλεγχο των μη κυβερνητικών οργανώσεων για την αξιολόγηση του έργου τους. Πάρα πολλέ μη κυβερνητικέ οργανώσει δραστηριοποιούνται αυτή τη στιγμή παγκοσμίω. Το έργο του κρίνεται από τα αποτελέσματα. Όμω, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα Εκτός από την οικονομική κρίση και τα επαχθή μέτρα που επιβάλλονται στους πολίτες από τους δανειστές, υπάρχει και το τεράστιο θέμα των μεταναστών που έχουν παραμείνει εγκλωβισμένοι στη χώρα μετά το κλείσιμο των συνόρων των ευρωπαϊκών κρατών. Εκεί έχουν βρει πρόσφορο έδαφος και δραστηριοποιούνται κάποιες μη κυβερνητικές οργανώσεις που ο ρόλος τους είναι ύποπτος και μπορώ να πω και επικίνδυνος. Κάποιοι υποτίθεται αλληλέγγυοι προσπαθούν να υποκαταστήσουν το κράτος. Δεν μιλάω για θέματα σύντησης και περίθαλψης κάποιες μη κυβερνητικές οργανώσεις υπονομεύουν την ίδια την ελληνική κυβέρνηση εκμεταλλευόμενη την απελπισία αυτών των ανθρώπων και διαδίδοντας ψεύδι και οδηγίες ότι θα ανοίξουν τα σύνορα χειραγωγούν και προτρέπουν σε αυτούς τους ανθρώπους να παραμείνουν κοντά στα σύνορα. Στην ειδωμένη όπου η κυβέρνηση προσπαθεί να απομακρύνει τους μετανάστες και να τους προωθήσει σε οργανωμένες δομές όπου θα έχουν ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης, κάποιες μη κυβερνητικές οργανώσεις παροτρύνουν τους μετανάστες να παραμείνουν εκεί με αποτέλεσμα να κινδυνεύει τόσο η υγεία τους αλλά και η ασφάλειά τους. 30 μέρες τώρα η σιδηροδρομική γραμμή της Ιδωμένης έχει καταληφθεί από μετανάστες με την παρότριση κάποιων ύποπτων μη κυβερνητικών οργανώσεων με αποτέλεσμα τεράστιο οικονομικό κόστος για την Ελλάδα. Για να ολοκληρώσω θα πρέπει, θα πρέπει πριν να χρηματοτηθούν κάποιες ΜΚΟ να εξεταστεί και ο ρόλος τους και τα αποτελέσματα του έργου τους. Σας ευχαριστώ. Ε, thank Σας ευχαριστώ. Και έτσι περνώ στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης, γιατί ο χρόνος μας εξαντλείται. Σας ευχαριστώ πολύ. Προθεσμία λοιπόν 21 Απριλίου, ψηφοφορία 15-16 Ιουνίου στην Επιτροπή, στην Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού τον Ιούλιο του 2016 και σας ευχαριστώ. Σημείο 11. Προετοιμασία της μετεκλογικής αναθεώρησης του πολίτου δημοσιονομικού πλησίου 2014-2020. Ο κύριος Πυρίνσκι έχει το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. όπως όλοι γνωρίζουμε, η μετεκλογική αναθεώρηση του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου είχε προβλεφθεί ως εργαλείο ώστε ο προπολογισμό της Ένωσης να προσαρμοστεί στις συνθήκες που ακολούθησαν την προσαρμογή του πλαισίου με τις νέες συνθήκες και βέβαια τις πολιτικές προτεραιότητες που θα είχε εντωμεταξύ ε, προωθήσει το Κοινοβούλιο, η Επιτροπή και το Συμβούλιο από κοινό. Η κατάσταση λοιπόν κατεπηγόντως και σαφέστατα πρέπει να προχωρήσει, είναι αναγκαία και το πολιτές οικονομικό πλαίσιο βρίσκεται σε ένα σημείο καμπής. Θα, λέναμε, θα λέγαμε, τα δημοσιονομικά μέσα έχουν σχεδόν εξαντληθεί και δεν έρονται στο ύψος των πολιτικών απαιτήσεων ακόμη και με την πλήρη ανάπτυξη των δυνατοτήτων που προσφέρει ευελιξία. Οι προκλήσεις λοιπόν που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση κατόπιν της υιοθέτησης του δημοσιονομικού πλαισίου σχετίζονται τόσο με την σαφή αδυναμία για επίτευξη των πιο σημαντικών προτεραιοτήτων της Ευρώπης 2020 και επιπλέον αυτού των απρόβλεπτων και μεγάλων προκλήσεων της ε, εισρωής ε, προσφύγων και όλα αυτά καθιστούν την αναθεώρηση του πολίτου δημοσιονομικού πλαισίου κατεπίγουσα και σημαντική ανάγκη. Οι στόχοι, όπως τους έχουμε για την Ευρώπη 2020, με 75% απασχόληση ε, για το 2020 είναι μακράν του να επιτευχθούν. Είμαστε στο 69% σήμερα. Ιδιαίτερα σοβαρά είναι τα προβλήματα για γυναίκε, ηλικιωμένου, άτομα με αναπηρίες νέου μενοτικές ομάδε. Και πιο ενισχυτικό απ' όλα, τα ποσοστά αύξηση τη μακροχρόνια ανεργία έχουν διπλασιαστεί από το 2,6 το 2008 το 5, ε, στο 5,1 το 2014. Και άρα το μερίδιο της μακροχρόνιας ανεργίας είναι ένα διαρκώς αυξανόμενο ποσοστό στα συνολικά ποσοστά της ανεργίας. Έχουμε επίσης πιεστικά και κατεπήγοντα προβλήματα με 4,4 εκατομμύρια νέους, 25%, ανεργ... 25 ε, εκατομμύρια συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2014 έχουμε μεγάλες προκλήσεις όπως είναι η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός που επίσης τα τελευταία χρόνια αυξάνονται με 5 εκατομμύρια επιπλέον στα 120 εκατομμύρια που είχαμε στην αρχή της περίοδου 24,4% κινδυνεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση από αποκλεισμό και φτώχεια. Ιδιαίτερα αυτό πλήττει τα παιδιά συνολικά ποσοστά 28% και σε ορισμένα κράτη-μέλη 50% ακόμη. 20 εκατομμύρια παιδιά δηλαδή ζουν σε οικογένειες που καθημερινά υποφέρουν από την απουσία εισοδήματος και βασικών υπηρεσιών, όπως στέγη, θέρμανση, τροφή, σχολείο, γιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Επίσης υπάρχουν οικογένειες με μειονοτικό ε, υπόβαθρο, ε, ιδιαίτερε δυσκολίες ε, και άλλες διτερότητες που βέβαια πάντα βαρύνουν ακόμη περισσότερο τα παιδιά. Πρέπει να κοιτάξουμε λοιπόν τις δυνατότητες της τάσης ευρωπαϊκής οικονομίας και ούτω καθεξής και είναι σημαντικό να εστιαστούμε στο εφικτόν αλλά ταυτόχρονα και να μην αποφύγουμε την προβολή μέτρων συγκεκριμένων επειδή θεωρούμε ότι να μην αρκέσουν οι πόροι. λοιπόν υπόψη και τελευταίων ε, δημοσκοπήσεων από ευρωπαϊκούς οργανισμούς που δείχνουν ότι 51% των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρούν ως κύρια προτεραιότητα την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού θα πρότεινα να εστιαστούμε προς το ελάχιστο απαραίτητο σε τρεις συγκεκριμένες αναθεωρήσεις. Πρώτον, το μερίδιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου να ανέρχεται στο 25% του συνολικού προπολογισμού συνοχής. Δεύτερον, να μην υπάρχουν περιορισμοί στις εθνικές πρικοδοτήσεις για το Κοινωνικό Ταμείο. Και τρίτον, να εξασφαλίζεται η ροή των πόρων για κάθε χρόνο. Επίσης, ένα δεύτερο κεφάλαιο θα πρέπει να υπάρχει ένα ειδικό ταμείο για την εξασφάλιση της ευρωπαϊκής εγγύησης παιδιών με ειδικούς πόρους, συγκεκριμένους πόρους, ώστε να βοηθηθούν και οι γονείς να αποφύγουν τον κοινωνικό αποκλεισμό και να εξασφαλίσουν μια θέση εργασίας. Η εγγύηση επίσης τρίτο κεφάλαιο για, τους, ναι, για την απασχόληση των νέων πρέπει να συνεχίσει να προσφέρεται τουλάχιστον στο 2020 και με σεβασμό των άρθρων του άρθρου 14 του πολίτου δημοσιονομικού σχεδίου. Οι αναμενόμενες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενόψη της αναθεώρησης του σου προκτάσης δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως ένα μέσο αντικατάστασης της απαραίτητης χρηματοδότησης ε, με στόχους ε, πολιτικούς. Τα μέτρα θα πρέπει να συνεχίσουν στην δρόμο της απλούστευσης και του συντονισμού μεταξύ των διαφόρων ταμείων, προκειμένου να εξασφαλιστούν καλύτερες επιδόσεις. Η αναθεώρηση του ποδοσού πάντως θα πρέπει να ορίσει νέες προτεραιότητες ανάλογα με τις κατεπίγουσες ανάγκες, νέες προτεραιότητες που θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο ποδοσού και η αναθεώρηση θα πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη ε, διαρκής και πάγιες ανάγκες που δεν έχουν αντιμετωπιστεί, απασχόληση κοινωνικά εν γέννη. Και πρόσθετη πόρη θα χρειαστούν καθώς οι υφιστάμενοι δεν αρκούν. Θα πρέπει επίσης να υπογραμμιστεί η ανάγκη αυτή η χρήση των υφισταμένων ε, μεσονομικών μέσων να μην οδηγεί σε συρρήγνωση του ευρωπαϊκού προπολογισμού γιατί αυτά τα μέσα είναι απαραίτητα για τις οικονομικές δραστηριότητες ε, και βέβαια θα έχουν χάρη στη χρηματοδότηση από τον Ευρωπαϊκό Προγραμματισμό σε συγκεκριμένου αντίκτυπο. Δεν θα πρέπει όμω να πηγαίνουν σε όλους τους τομείς πολιτική καθώ υπάρχουν τομεί. Όπου ακριβώ μπορεί η δημόσια χρηματοδότηση να φέρει αποτελέσματα. ενώ η ειδική χρηματοδότηση μπορεί να μην τα καταφέρει. Και έχουμε νομίζω πρόεδρε σημαντική δουλειά να κάνουμε. Είναι μια γνωμοδότηση η οποία θα προσφέρει ουσιαστικά στην Επιτροπή των Προπολογισμών και την τοποθέτησή της που θα είναι η θέση του Κοινοβουλίου. Και γι' αυτό περιμένω να συνεργαστούμε με τους και και να ακούσω τις προτάσεις τους. για να έχουμε μια καλή θέση. Και ευχαριστώ. Thank you, Mr. Σας ευχαριστώ. Ο σκιωδής του ΕΛΚ παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον κύριο Περινσκή για την ε, δουλειά που έχει γίνει που έχω την εντύπωση ότι είναι μια πολύ καλή βάση δουλειάς και ε, νομίζω ότι θα μπορέσουμε να επιτύχουμε συμβαστικές λύσεις. Ε, δεν θέλω να φαίνομαι υπερβολικά αισιόδοξο, αλλά νομίζω ότι θα καταφέρουμε να βρούμε λύση. Και εδώ πρέπει να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση που αντιμετωπίζουμε σήμερα ως Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με τα θέματα προϋπολογισμού και ε, περιορισμού των χρηματοδοτήσεων ε, εν ώψη του ορίζοντα 2020 τα περισσότερα από τα ανώτατα όρια έχουν ήδη ξεπεραστεί λόγω μια σειρά από προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφέρεται η γνωμοδότηση στην ανάγκη επενδύσεων, αυτό δεν μπορούμε παρά να το υπογραμμίσουμε και επίσης η πρωτοβουλία του ε, επενδυτικού ταμείου ε, είναι απολύτως ε, θετική. Και σκέπτομαι τις επιτυχίες ε, του αναπρογραμματισμού ως προς τον ορίζοντα 2020 και θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω τη σημασία του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Γνωρίζουμε ότι σήμερα το Ταμείο υφίσταται πιέσεις και αντιμετωπίζει διάφορες προκλήσεις ώστε να δώσει απαντήσεις στα προβλήματα ε, σχετικά με τους ε, πρόσφυγες. Αλλά αυτά τα νέα προβλήματα ε, δεν πρέπει να μας απομακρύνουν από τον αρχικό μας στόχο γιατί θα πρέπει να δούμε, να εξετάσουμε εκείνες τις κοινωνικές κατηγορίες του πληθυσμού που είναι οι περισσότερο ευάλωτες, οι περισσότερο εκτεθειμένες. Θα πρέπει επίσης ε, να έχουμε ιδιαίτερη προσοχή ε, ε, στην ανάπτυξη μηχανισμών εκμάθησης και κατάρτισης που είναι πολύ σημαντικό στοιχείο στα πλαίσια της απασχόλησης. Αυτά είναι τα στοιχεία που αυτή τη στιγμή μας φαίνονται ε, ουσιώδη και σε κάθε περίπτωση ο εισηγητής μπορεί να βασίζεται στην δική μας υποστήριξη ώστε να έχουμε ένα κείμενο όσο πιο συνενετικό γίνεται αλλά όσο και πιο περιεκτικό. Επιτρέψτε μου μία παρατήρηση προσωπική εδώ είναι σημαντικό να εργαζόμαστε στην αναθεώρηση, αλλά ε, προσωπικά πιστεύω ότι δεν θα μπορέσουμε ποτέ να ξεπεράσουμε το πρόβλημα αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον δεν έχουμε έναν προϋπολογισμό αξιοπρεπή. Γιατί στα επίπεδα που έχουμε φτάσει πρέπει να είμαστε σοβαροί και να το αναγνωρίζουμε, δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειαζόμαστε ίδιους πόρους για να καλύψουμε τα ζητήματα αυτά και να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον ε, εισηγητή για τη δουλειά του. Οι προτάσεις του συνιστούν καλή βάση για τη συζήτηση για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί τη βάση των θεμάτων ε, της, ε, των κοινωνικών και της ε, εργασίας. Βεβαίως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αντιμετωπίσει λόγω και της μεγάλης οικονομικής κρίσης προβλήματα ανεργίας σοβαρά οι δυνατότητες του προπολογισμού έχουν σχεδόν εξαντληθεί τα τελευταία δύο χρόνια. Έχουν γίνει μεγάλες προσπάθειες για απορρόφηση κονδυλίων. Τώρα υπάρχει ωστόσο ανάγκη να εξασφαλιστεί ένα περιθώριο για διαχείριση των νέων προβλημάτων. Και όπως είπε και ο συνάδελφος, σε ένα βαθμό υπάρχει ε, υπάρχουν όλα αυτά τα προβλήματα που μας εξέθεσε. Υπάρχει ωστόσο και το ζήτημα της μετανάστευσης με κόστος δισεκατομμύρια, εσωτερικά προβλήματα ασφάλειας, προβλήματα στη γεωργία λόγω των κυρώσεων της Ρωσίας, τα ανεπίλητα ζητήματα των ε, υπερβολικά υψηλών αναλήψεων υποχρεώσεων του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι λοιπόν ε, ένα δημοσιονομικό πλαίσιο το οποίο έχει διατυπωθεί κατά τρόπο ε, πολύ ανελαστικό και επίση πριν από μεγάλο διάστημα και άρα δεν μπορεί να προσαρμοστεί στι νέε συνθήκε, σημαίνει ότι θα πρέπει να διατυπώσουμε εμεί νέε προποθέσει. Ε, χρειάζεται δηλαδή να ενισχυθεί ο προπολογισμό, αλλά δεδομένων των γενικών οικονομικών συνθήκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το αίτημα δεν μπορεί να προβληθεί. Χρειάζεται λοιπόν, γιατί θα χρειαζόντουσαν επιπλέον φόροι και θα έπρεπε βέβαια να έχουμε υπόψη ότι ο πολίτη ε, μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα τα, τα χρήματά του από ότι ο πολιτικό στη θέση του. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να αποφύγουμε περαιτέρω ανελαστική χρήση. Η χρήση των κονδύλιων θα πρέπει να ε, επαληθεύεται πολύ πιο αποτελεσματικά και να είναι καλύτερη και πιο αποτελεσματική αυτή η χρήση. Ε, θα πρέπει να ανθαρρύνεται η καινοτομία, οι επιστήμες, η αρχή της προστιθέμενης αξίας, μία από τις πέντε αξίες ε, για την κατάρτιση του προπολογισμού από το 2010, σημαίνει ταυτόχρονα και πιο αποτελεσματική διαχείριση του προπολογισμού, δηλαδή σε επίπεδο εθνικό στο δυνατόν περισσότερο, γιατί έχει ο πολίτης το δικαίωμα να ε, εξασφαλίζει την προσεκτική και συνετή διαχείριση των χρημάτων του και γι' αυτό πρέπει πάντα να επαληθεύεται κάθε μέτρο και εκτέλεσή του πριν να διατίθεται πεστρά κονδύλια. Η εγγύηση για την ενεργεία των νέων, ειναι παραδείγματι, υπάρχουν κράτη-μέλη τα οποία δεν μπόρεσαν να υλοποιήσουν κατά τρόπο αποτελεσματικό σε διοικητικό επίπεδο τα μέτρα που προβλέπεται. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται μια αξιολόγηση προτού να διατεθούν περαιτέρω μέσα. Επιπλέον θα πρέπει να καταστήσουμε απολύτω ε, σαφέ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα χρήματά τη δεν μπορούν να, να αντικαθιστούν εθνικά προγράμματα. Μπορούν να τα συμπληρώσουν ναι. Και αυτά βέβαια με βάση και τις απαιτήσει που έχει προσδιορίσει για την αποτελεσματική διαχείριση του προπολογισμού η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να κοιτάξουμε σε ποιου τομεί θα πρέπει να γίνουν οι περικοπέ των κονδυλίων για να εξασφαλιστεί μια καλή ισορροπία στον προπολογισμό. Παρακαλώ οι πάντε να αναλογιστούν ποιε πρέπει να είναι οι προτεραιότητέ μα και αν είναι διατεθειμένοι να ε, ε, παρετηθούν από αιτήματα και προτιμήσεις ε, που, έχουν, που έχουμε όλοι διατυπώσει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Χάρκιν Σκιώτης για την Άλτα. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω λοιπόν για μια πολύ καλή γνωμοδότηση η οποία συνιστά την σωστή βάση ε, από την οποία να ξεκινήσουμε τις διαβουλεύσεις μας. Στόχος της αναθεώρησης αυτής είναι να καταστήσει ικανό το Κοινοβούλιο να επανεξετάσει τις προτεραιότητες του υπό το φως των αλλαγών που έχουν συμβεί εν τω μεταξύ. Ιδιαίτερα βλέποντας για την οικονομική κατάσταση και τις μακροοικονομικές ε, ε, προβλέψεις δεδομένα. Θα συμφωνήσω ότι το MFF είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση και όταν βλέπουμε τις νέες προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζουμε και που εμφανίστηκαν τα τελευταία τρία χρόνια, αναφερθήκατε ήδη στο θέμα των προσφύγων, της κρίσης των προσφύγων. Υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί. Ανεργία, όχι μόνο ανεργία, αλλά μακροπρόθεσμη ανεργία. Αύξηση της φτώχειας, αύξηση της φτώχειας που χτυπάει ιδιαίτερα τα παιδιά, που έχει τεράστιες μελλοντικές επιπτώσεις και στον τομέα της κατοικίας και της υγείας και της εκπαίδευσης η κάλυψη, η, μάλλον οι ευθύνε μας σε σχέση με τους αναπήρους επί τη βάση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών. Βλέπουμε ότι έχουμε τεράστια προβλήματα, ήταν ήδη μεγάλα τα προβλήματα για τον προϋπολογισμό και τώρα έχουμε επιπλέον. Θα συμφωνήσω λοιπόν ότι αυτά τα οποία αποφασίζουμε θα πρέπει να είναι εφικτά, αλλά δεν έχουμε τους πόρους έχουν εξαντληθεί δυνατότητες και πώς μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι αυτά τα οποία αποφασίζουμε θα γίνουν εφόσον δεν έχουμε τους απαιτούμενους πόρους. Δεν ξεκινάμε από το μηδέν βέβαια. Υπάρχουν έτσι και λιώς εθνικές παρεμβάσεις, υπάρχουν ε, άλλα μέσα όπως η πολιτική συνοχή, τα διαφθρωτικά ταμεία, έχουμε νομικές υποχρεώσεις έχουμε ευθύνε και σε σχέση με το ΠΔΠ για να πετύχουμε τους στόχους μας. Ξέρουμε όμως ότι τα όρια έχουν εξαντληθεί και οι δυσκολίες είναι πολλές. Θα συμφωνήσω λοιπόν με τον εισηγητή ότι πρέπει να επανεξετάσουμε τις πολιτικές μας προτεραιότητες. Δεν μπορούμε να προσθέτουμε στόχους και αυτό που κάνουμε σήμερα είναι να ελέγξουμε το ποιες είναι οι προτεραιότητες αυτές και είναι αλήθεια ότι όλοι μας θα θέλαμε να έχουμε ένα μακρότατο κατάλογο, αλλά παρόλα αυτά μόνο στην περίπτωση που έχουμε τους απαιτούμενους πόρους. Πρέπει να είμαστε ευέλικτοι, αλλά ταυτόχρονα και ιδιαίτερα πειθαρχικοί. Δεν έχει σημασία από ποια πολιτική ομάδα καταγόμαστε, αλλά κανένας δεν μπορεί να αγνοήσει τη σοβαρότητα του προβλήματος των προσφύγων στην παρούσα φάση. Συζητάμε λοιπόν τα θέματα αυτά για τις προτεραιότητές μας και στην δική μας πολιτική ομάδα. Οι πρωτοβουλίες για την απασχόληση των νέων είναι πάρα πολύ σημαντικές, αλλά σύμφωνα με το Διεθνής Γραφείο Εργασίας η εγγύηση για την απασχόληση των νέων είναι υποχρηματοδοτούμενη κατά ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό. Κάποια τελικά σχόλια τώρα για την ε, παιδική εργασία και θα πρέπει, ή μάλλον για την φτώχεια και το πώς χτυπά τα παιδιά. Όταν βλέπει τα στοιχεία κανείς για τους ε, για τα ορφανά παιδιά, για τα παιδιά με αναπηρίες, για τα παιδιά θύματα σωματεμπορίας, για τα παιδιά των προσφύγων. Ο αριθμός μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερος και ποιος ε, μπορεί να είναι κατά της λήψης μέτρων προς την κατεύθυνση αυτή. Από την άλλη, εάν δεν έχουμε την απαιτούμενη ευελιξία για να πάρουμε τα σωστά μέτρα και σε δημοσιονομικό επίπεδο, θα πρέπει να ξέρουμε που ε, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί μια τέτοια εγγύηση για τα παιδιά, αλλά θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, να μην υποσχόμεθα πράγματα που δεν μπορούμε να παραδώσουμε. Ίσως θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι σε αρκτικό επίπεδο, δεν λέω όχι, αλλά έχουμε την ευθύνη να είμαστε σίγουροι ότι αυτό το οποίο θέλουμε να πετύχουμε είναι εφικτό και το είπε και ο εισηγητής. Λοιπόν, είναι τεράστιο το πρόγραμμα αυτό, είναι πολύ σημαντικό και θα πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας έτσι ώστε να καλύψουμε τις προτεραιότητές μας πολιτικά ακόμα και αν κάτι τέτοιο μερικές φορές είναι πραγματικά δύσκολο. Πάντως είναι πολύ σημαντικό το σχέδιο αυτό και θα το στηρίξω. Ευχαριστώ. Σκιώδη Σκιώδης της Γκουε δεν είναι εδώ. Λόπες όχι. Για τους πράσινους. Ευχαριστώ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Και ευχαριστώ και τον εισηγητή για μια πολύ καλή και ισορροπημένη γνωμοδότηση που είναι πολύ καλή βάση να εργαστούμε. Εμείς ε, θα εστιαστούμε σε τρία σημεία στροπολογίες μας. Η αναθεώρηση των ανώτατων ορίων του MFF. Δεύτερον, ότι ο ροϊκός προϋπολογισμός θα πρέπει να καλύπτει τους κοινωνικούς στόχους του 2020. Και τρίτον, το ESF και το 20% του ESF το οποίο αποσκοπεί την κοινωνική συνοχή. Χρειάζεται ανάπτυξη ε, δεξιοτήτων και κατάρτιση συμπεριλαμβανομένων πράσινων θέσεων απασχόλησης. Αυτό, αυτά από πλευράς μας ε, περιμένουμε με ενδιαφέρον τη συζήτηση και την ανάπτυξη της κοινή μας θέσης. ε, του Ιευθυντή, παρακαλώ. Ε, σας ευχαριστώ. Εγώ παρακολουθώ τις εργασίες αυτές ε, για την ε, ΛΥΜΠΕ επίσης και είναι πολύ σημαντικό που μπορώ να έχω αυτήν την διπλή διάσταση και τη διπλή οπτική γωνία. σχετικά με τους ε, πόρους που χρειαζόμαστε και μας λείπουν, είτε θα πρέπει να τους βγάλουμε από κάποιο μαγικό καπέλο, γιατί είδα ότι καταφέραμε να δώσουμε 3 δισεκατομμύρια στην Τουρκία για τους ε, Σύριους πρόσφυγες. Αλλά όταν χρειάζεται να μαζέψουμε κάποιους πόρους για σοβαρά κοινωνικά προβλήματα, ξαφνικά ανακύπτουν εμπόδια. Λέω λοιπόν ότι εφόσον βρήκαμε τρία δις για να δώσουμε στην Τουρκία, πρέπει απαραίτητο να βρούμε πόρους για τα προγράμματα που υποστηρίζουν την Ευρώπη μας και την κοινωνική της διάσταση. Προφανώς και θα πρέπει αλληλέγγυα να αντιμετωπίσουμε και το πρόβλημα των μεταναστών, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Εμείς, ε, μάλλον ο πρόεδρος Γιούνκερ, ε, δημιούργησε αυτό το... Ε, στα πλαίσια του, του, των μεγαλόπνων δηλώσεων του δημιούργησε ένα, θα έλεγα, φαντασματικό ε, οικοδόμημα χρηματοδότησης που τελικά δεν υπήρχε αλλά στην πραγματικότητα αφαίρεσε σημαντικούς πόρους από πραγματικά προγράμματα τα οποία έτρεχαν και τα οποία είχαν μεγάλη χρησιμότητα γιατί χρηματοδοτούσαν την έρευνα και την ανάπτυξη. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο μπορούμε να κάνουμε. Δηλαδή έχουμε προγράμματα που δεν είναι φανταστικά, δεν είναι φαντασιώσεις, είναι πραγματικά προγράμματα και αντιμετωπίζουν την ανεργία και τα κοινωνικά προβλήματα και από εκεί αφαιρούμε πόρος για να χρηματοδοτήσουμε τεράστια έργα και τεράστιες επενδύσεις οι οποίες τελικά δεν οδηγούν στην δημιουργία θέσεων απασχόλησης αυτά τα τεράστια έργα υποδομής γιατί μπορεί να φτιάξεις ένα αυτοκινητόδρομο ο οποίος δεν χρειάζεται πολύ μεγάλη συντήρηση πέραν του γεγονότος ότι έχει καταστρέψει την Ήπεθρο ούτε οδηγεί σε μόνιμες θέσεις απασχόλησης. Εγώ γνωρίζω ότι η δημιουργία ενός ταμείου υποστήριξης των παιδιών σήμερα φαίνεται αδύνατον. Αλλά έχουμε ένα εκατομμύριο παιδιά στην Ευρώπη που υποφέρουν από υποσιτισμό στην ουσία και κακής ποιότητας διατροφή. Θέλουμε να το δούμε αυτό το πρόβλημα. Ή θα πρέπει να λειτουργήσουμε κι εμείς ως άλλη μια χώρα από αυτές που θα, που θα είναι κατάλληλες ως προορισμός βοήθειας κοινωνικής. Θα πρέπει να επενδύσουμε, θα πρέπει να βρούμε τους πόρους. Γιατί αυτή η αναθεώρηση το μόνο σαφές μήνυμα που διαβιβάζει είναι ότι Έχουμε φτάσει στα μισά του δρόμου και έχουν τελειώσει τα λεφτά. Όλα τα προγράμματα ασύλου και μετανάστευσης τελείωσαν οι πόροι. Τα προγράμματα του Κοινωνικού Ταμείου για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού απολυσμού τελείωσαν και είμαστε στα μισά του δρόμου. Τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή, άλματα πίστεως, να βάλουμε τα κλάματα, δεν έχουμε πια λεφτά, τι θα κάνουμε, τι πρέπει να κάνουμε πρέπει να κάνουμε να προχωρήσουμε σε θαραλέες αποφάσεις και επιλογές. Έχουμε το πρόβλημα της μετανάστευσης που καλούμαστε να το διαχειριστούμε. Έχουμε το πρόβλημα της φτώχειας στην Ευρώπη. Στην Ιταλία, στη χώρα μου, έχουμε 7 εκατομμύρια που δεν αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της φτώχειας, ζουν στη φτώχεια. Δεν, τα, όρια, τα όρια που κάποτε συζητούσαμε δεν είναι πραγματικά. Η κατάσταση είναι χειρότερη και αυτή η κατάσταση είναι απόλυτης προτεραιότητας. Η δική μας στήριξη θα είναι απόλυτη στην γνωμοδότησή σας. Αλλά αν βγάλετε το Ταμείο Εγγύησης για τα παιδιά, εμείς δεν θα μπορέσουμε αυτό να μην το ε, σημειώσουμε, διότι δεν γίνεται να μην φροντίσουμε τα παιδιά μας. Ευχαριστώ. Κύριε Μπιζωτό δεν είναι εδώ. Κύριε Δομινίκη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ανακοιγνώσκω τις ε, σκέψεις της κυρίας Μπιζωτό. Η μετεκλογική αναθεώρηση του πολίτου δημοσιονομικού σχεδίου θα πρέπει να λαμβάνει καλύτερα υπόψη την ανικανότητα των κρατών μελών για αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων ή διαρκής επαναγραφή σε περίπτωση Κάτι κατεπίγουσων αναγκών ε, για τις στρατηγικές ε, διαρθρωτικής ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, σε αιτήματα για νέες αυξήσεις στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ε, είναι οι συνέπειες αυτών των που, θα πρέπει επιπλέον να πληρώσουν και να έχουν ήδη γονατίσει από την οικονομική κρίση οι πολίτες μας τα χρήματα αυτά που συνεχίσουν να αποτελούν διασπάθηση πόρων το 2015 τον Απρίλιο είχαμε 28 εκατομμύρια, 4,5 συγκεκριμένα νέοι κατά τον 25 άνεργοι. Ε, έτσι λοιπόν αυτή είναι η στρατηγική της Ευρώπης 2020 για να εξασφαλιστεί η ανάπτυξη με συγκεκριμένα και αποτελεσματικά ε, μέσα χωρίς διασπάθηση χρήματος αντιμετώπιση των προβλημάτων της εργασίας θα έπρεπε πρώτον να υποστηρίζονται και να διδονται προτεραιότητες στα κράτη-μέλη. Δεύτερον, να προσφέρονται πρωτοβουλίες όχι μόνο για την προσφορά στην εργασία αλλά και στη ζήτηση. Και τρίτον, να ενισχύεται κάθε έργο το οποίο στόχο θα έχει να ε, ενισχύει την κατάρτιση στην επιχείρηση. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ. Η κυρία Σάρτια. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να πω στον συνάδελφο κύριο Πυρίνσκι πόσο ενδιαφέρουσα είναι η δουλειά του, πόσο πολύ αξίζει να την υποστηρίξουμε και για διάφορους λόγους. Καταρχάς γιατί ο Ζαν Κλοντ Juncker όταν ήρθε να μας μιλήσει μίλησε για τριπλό αλφα στην ε, κοινωνική Ευρώπη και είπε ότι, αυτή, ότι η, επιτροπή μας, η Επιτροπή Εκτελεστική θα ήταν ε, αυτή τη φορά ε, κοινωνική επιτροπή. Έχουμε βαρεθεί λοιπόν να ακούμε επιχειρήματα που στηρίζονται μόνο σε δημοσιονομικού όρου. Η Επιτροπή Απασχόληση δεν μπορεί να κοιτάει μόνο ε, τα προβλήματα σε όρου προπολογισμού. Εμείς θέλαμε συγκεκριμένε πολιτικές κατευθύνσεις, συγκεκριμένους πολιτικούς προσανατολισμού ε, προβάλλουμε και απαιτούμε και γι' αυτό και σε αυτό συμφωνώ με τον εισηγητή και την πλειοψηφία των σκιωδών. Το είπε η κυρία Χαρκίνο ότι βρισκόμαστε σε ένα σημείο καμπής, ε, έχουμε να κάνουμε οικονομικές πιέσεις αφόρητες αυτή τη στιγμή και χρειάζεται όχι τόσο πολύ θάρρος όσο αιμονή και επιμονή με, τις, με τα νέα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, τις νέες προκλήσεις και δι απασχόληση και μετανάστες, θα πρέπει όλο και περισσότερο να εμένουμε με σταθερότητα στη διεκδίκηση των κοινωνικών πολιτικών που θέλουμε. Εγώ λοιπόν επιμένω σε πέντε σημεία συγκεκριμένα. Το πρώτο και πολύ σωστά επισημαίνεται στην έκθεση. 13,1% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης διατίθεται για τη διάσταση των τραπεζών και μόνο 1% για τις ε, πολιτικές που στόχο έχουν να υποστηρίξουν την απασχόληση και τις πολιτικές της συνοχής. Επομένως, ναι, πρέπει να είμαστε άτεγκτοι στην υπόθεση αυτή. Δεύτερον, η απασχόληση έχει θεμελιώδη σημασία και αξία. Δεν θα ήθελα, υπό το φως μιας αναθεώρησης, επί τη ευκαιρία μιας αναθεώρησης, να ανατραπούν τα ιερά και όσια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου δεν μπορούμε να συγχωνεύσουμε το κοινωνικό ταμείο που στόχο έχει την, τη στήριξη στην απασχόληση με ταμεία συνοχής. Πρέπει λοιπόν να παραμείνει στο πυρόβλητο το κοινωνικό ταμείο και αυτό είναι απαραίτητο και επιπλέον, για να αναφερθώ και στην τρίτη, στο τρίτο επιχείρημα, θα χρειαστεί και για να αντιμετωπιστεί η μετανάστευση υπό το φως αυτής της αναθεώρησης και επί τη ευκαιρία της αναθεώρησης να περάσουμε στο 25% του Ταμείου Συνοχής για το Κοινωνικό Ταμείο. Απαραίτητο. Τέταρτο. Όχι, μάλλον στα 25% πρέπει να διαφυλαχθούν τα 20% για την καταπολέμηση της ε, φτώχειας. Αυτά είναι απαραίτητα. Ύστερα από τα όσα ακούσαμε για τη φτώχεια και κυρίως τη φτώχεια των παιδιών. Τέταρτον, πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων. Πολλέ φορέ έχω λάβει το θέμα, στο θέμα αυτό το λόγο, κυρία Πρόεδρε, και στο συγγνώμη που επανέρχομαι. Αλλά η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων οδήγησε σε σημαντικές συγχύσεις, πιστεύω, παρερμηνίε σε επίπεδο κρατών μελών και οι υπουργοί ακόμη δεν ξέρουν τι ακριβώ συμβαίνει και σημαίνει. Ενδιαφέρον λοιπόν θα ήταν μόνο το θέμα της ενίσχυσης αυτής της πρωτοβουλίας στις πιο δύναμες ε, οικονομικά περιοχές. Απέκλειπτο όμως και την ουσία της πολιτικής μας που είναι η εγγύηση για την νεολαία. Πρέπει λοιπόν να επανέλθουμε και να προβάλλουμε ιδιαίτερα την εγγύηση για την νεολαία. Τελευταίο, ας μην ε, την πατήσουμε τα λειτουργικά προγράμματα σε κάθε κράτος ύπογραφηκαν κατά, με μεγάλες καθυστερήσεις. Έτσι λοιπόν δεν μπορούμε να έχουμε μόνο ποσοτικές αξιολογήσεις γιατί αλλιώς καταστρέφονται όλα τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολιτικά εμείς έχουμε δίκιο. Πολιτικά η δική μας η γραμμή, η γραμμή της Επιτροπής Επασχόλησης είναι η γραμμή που θα πρέπει να επικρατήσει. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Πυρίνσκι για την γνωμοδότησή του. Είναι δύσκολο να μην συμφωνήσει κανείς με αυτά τα οποία λέγει η πρότασή του. Και σχετικά με την συνέχιση της ε, πρωτοβουλίας αυτής. Αυτός ο τομέας τον οποίο καλύπτει η πρόταση είναι ένας πάρα πολύ ευαίσθητος τομέας ε, και πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας και τον ευχαριστώ πολύ. Έχοντας ακούσει τώρα τις συζητήσεις οι οποίες προηγήθηκαν, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε κάτι το οποίο δεν βρίσκω στην έκθεση αυτή. Θα ήθελα να υπάρξει ειδική προσοχή σε θέματα συντονισμού των μεμονωμένων διαφθορτικών ταμείων ανάμεσα σε προγράμματα τα οποία είναι στη διάθεσή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν πράγματι στρέψουμε την προσοχή μας εμείς στη γνωμοδότηση αυτή και ζητήσουμε την αύξηση των δημοσίων επενδύσεων, αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει νέες θέσεις απασχόλησης. Νομίζω ότι χωρίς την αύξηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου αυτό θα ήταν δυνατόν εφόσον υπάρξει καλύτερος συντονισμός ανάμεσα στο Περιφερειακό Ταμείο και το Νέο Ταμείο για Επενδύσεις. σαν παράδειγμα η υποστήριξη των επιχειρηματιών να δημιουργήσουν νέες θέσεις απασχόλησης, εάν πράγματι μπορούν να δημιουργήσουν τέτοιου είδους θέσεις, τότε πράγματι το διαφορετικά ταμεία, τα διαφορετικά ταμεία θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν αποτελεσματικά. Συνεπώς, θα ήθελα να σας ζητήσω να σκεφτούμε για μια ακόμη φορά τον συντονισμό των διαφορετικών ταμείων τα μέσα τα οποία έχουμε μέχρι τώρα στη διάθεσή μας είναι ανεπαρκή και δεν μπορούν να, να λειτουργήσουν αποτελεσματικά. Ευχαριστώ. Για Σλοβιέσκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η προσπάθεια δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να επιδιώξουμε. Και όπως είπε η Ελίζαμπεθ, θα πρέπει στο μέλλον το κοινωνικό ταμείο να είναι τουλάχιστον στο επίπεδο του 25% προορισμένο για την καταπολέμηση της φτώχειας. Αυτό ίσως ε, να μην είναι βέβαια στην εποχή μας ε, ε, επαρκές γιατί θα πρέπει να καλύψουμε όλες τις κοινωνικές κατηγορίες και διαστρωματώσεις και τους νέους και τους πλέον ηλικιωμένους και στόχος μας είναι να προετοιμάσουμε ένα πλαίσιο το οποίο να είναι πρόσφορο ε, για την προσαρμογή των Ευρωπαίων στην ψηφιοποίηση. Γι' αυτό λοιπόν ίσως και ένα 30% να ήταν καλύτερο. Στα πλαίσια της πολιτικής συνοχής όλο και περισσότερες περιοχές, περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχουν κάποια χαρακτηριστικά που θα τα χαρακτηρίζουν ακριβώς σαν χώρες προχωρημένες, προοδευμένες, κάτι το οποίο θα αποκλείει τις χώρες μας, ορισμένες τουλάχιστον από αυτές, από επιδοτήσεις που θα μας προετοιμάσουν καλύτερα στην για, για τον χώρο της εργασίας. Η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύντομα παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Ήταν πολύ ενδιαφέρον να παρακολουθήσει κανείς τη συζήτηση σήμερα. Ευχαριστώ τα μέλη της Επιτροπής σας. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία στα πλαίσια της αναθεώρησης του MFF να θεωρήσουμε ότι έχουμε μια ευκαιρία για τη βελτίωση των κοινωνικών μας πολιτικών και της παρέμβασης στον κοινωνικό τομέα. Προετοιμαζόμενοι και για την περίοδο μετά το 2020. Έχω την αίσθηση ότι τελευταία αυτή η γνωμοδότηση θα είναι σημαντική για μας για να προετοιμαστούμε σωστά, τίποτα περισσότερο. Σας ευχαριστώ. Ο κ. Σπυρίνσκι για να κλείσει η συζήτηση. Εγώ εκτιμώ ιδιαιτέρως τις αντιδράσεις των συναδέλφων Θα συμφωνήσω επίσης και με την υπογράμμιση από πλευρά σας των προτεραιοτήτων των πολιτικών τις οποίες έχουμε και του σεβασμού συγκεκριμένων κατά προτεραιότητα στόχων. Εφόσον είμαστε σοβαροί στα πλαίσια της αναγνώρισης της φύσης του προβλήματος, ζούμε μια περίοδο θα έλεγα ιδιαίτερα δύσκολη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ακραία δύσκολη, και υπάρχουν παρόλα αυτά οι προσδοκίες ότι κάτω από τέτοιες συνθήκες η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να παίξει έναν ορατό και ισχυρό ρόλο για τους πολίτες και από τους πολίτες. Ταυτόχρονα θα πρέπει να παραμείνουμε αρκετά συντηρητικοί θα έλεγα λέγοντας ότι η κατάσταση είναι αυτή όπως τη βλέπουμε και βλέπουμε και ποια είναι και τα όρια. Σε αυτή την περίπτωση αν είμαστε απλά παθητικοί και διαπιστώνουμε τα πράγματα τότε δεν θα έχουμε φέρει σπέρα στην υποχρεωσή μας. Βέβαια το εφικτό δεν θα πρέπει να το αγνοήσουμε. Όταν όμως ότι κατανοούμε ότι θα πρέπει να δοθούν προς την Τουρκία τρία δις μέσα σε λίγες εβδομάδες και αυτό από ό,τι φαίνεται είναι εφικτό, δεν νομίζω ότι θα πρέπει να αγνοήσουμε από πλευράς μας την πραγματική ανάγκη η οποία υπάρχει για άμεση δράση στους τομείς τους οποίους προανέφερα. Έγιναν και κάποιες κριτικές για καλύτερο συγχρονισμό ανάμεσα στις διαφορετικές μορφές χρηματοδότησης. Νομίζω λοιπόν ότι η σωστή χρήση των πιστώσεων είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να λειτουργήσει με αποτελεσματικό τρόπο και θα εκτιμούσα ιδιαιτέρως οι προτάσεις σας να κατατεθούν και οι τροπολογίες σας και να μπορέσουμε να τις εξετάσουμε από κοινού, καταλήγοντας σε μία θέση της Επιτροπής Απασχόλησης, που όπως είπε η κυρία Σούκοβα, θα εντάσσεται σε ένα σύνολο προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που να αναγνωρίζει το τι αναμένεται από αυτήν την αναθεώρηση, την ενδιάμεση και ταυτόχρονα και σαν Κοινοβούλιο και σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσπαθήσουμε να πετύχουμε τον στόχο αντιμετώπισης αυτών των σχετικά πρόσφατων αλλά και ιδιαίτερως πρόσφατων και σοβαρών προκλήσεων. Σας ευχαριστώ όλους. Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών 22 Απριλίου, 12η Μεσημβρινή, ψηφοφορία 24 Μαΐου, στην Επιτροπή Προϋπολογισμών 15-16 Ιουνίου και ελπίζω να φτάσουμε στην Ολομέλεια τον Ιούλιο. Σας ευχαριστώ. Τώρα θα γίνει μια παρουσίαση μιας μελέτης την οποία εμείς παραγγείλαμε για το πώς η απασχόληση και τα κοινωνικά θέματα αντιμετωπίζονται στα πλαίσια του Μηχανισμού Διακυβέρνησης του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και της συνεισφοράς των κοινωνικών δικτών που εφαρμόζονται στις μακροοικονομικές προβλέψεις από το 2013. Δεν είμαστε πάρα πολλοί, αλλά έχω την αίσθηση ότι μπορούμε και ίσως κάποιοι από εσά μπορούν να ακούνε τη συζήτηση και από τα γραφεία του. Στη Μανουέλα Λοντοβίτσι λοιπόν, από το Ινστιτούτο Κοινωνικής Έρευνας της Ιταλίας, θα κάνει μια ελπίζω συνοπτική παρουσίαση και ελπίζω να μείνουν και λίγα λεπτά για ερωταπαντήσεις. Έχετε το λόγο κυρία Λοντοβίτσι. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση για να παρουσιάσουμε αυτή τη μελέτη που κάναμε πέρυσι. Είμαστε ένα Ινστιτούτο Κοινωνικής Έρευνας με έδρα στην Ιταλία η κύρια εστίαση της μελέτης αυτής είναι πώς η απασχόληση και τα κοινωνικά ζητήματα καλύφθηκαν από το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο από το 2011. Ποια υπήρξε η συνεισφορά των κοινωνικών δικτών ή στη διαδικασία της μακροοικονομικής εποπτείας από το 2013 και ποιοι είναι η άποψη και η εντύπωση για τη διαδικασία που έχουν οι πιο σημαντικοί ενδιαφερόμενοι φορείς. Η μελέτη βασίστηκε στην εξέταση της νομοθεσίας και των σχετικών εγγράφων, αλλά και σε μια μελέτη πεδίου με 46 ενδιαφερόμενες φορείς σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Είχαμε συνεντεύξεις και τηλεφωνικές επαφές και συνεντεύξεις με εκπροσώπους ευρωπαϊκών φορέων και εθνικών φορέων και κάναμε και μία ενδελεχή αξιολόγηση οκτώ χωρών που είναι αντιπροσωπευτικές των διαφορών κοινωνικών συνθήκων που ισχύουν στην Ευρώπη. Όλα αυτά βρίσκονται στην περιγραφή και στα πορίσματα της μελέτης. Προτού παρουσιάσω τα κυρίως πορίσματα, θα άξιζε να πω δύο λόγια για το ευρωπαϊκό εξάμεινο, γιατί πρόκειται για μια περίπλοκη διαδικασία συντονισμού που ετέθησε εφαρμογή το 2011, όπως είπα, προκειμένου να συντονίσει δύο πολύ διαφορετικούς μηχανισμούς διακυβέρνησης των, ε, εκείνων την, της μακροοικονομικής εποπτείας επί τη βάση συγκεκριμένων διατάξεων της νομοθεσίας σχετικά με μακροοικονομικές ανισορροπίες που παρουσιάζουν συγκεκριμένες ε, χώρες του Συμφώνου Σταθερότητας αλλά και του συντονισμού του μηχανισμού κοινωνικής πολιτικής και απασχόλησης που βασίζεται στην ανοιχτή μέθοδο συντονισμού η οποία δίνει πολύ περισσότερο περιθώριο ευελιξίας στα τη μέλη να παρακολουθούν τους δικούς τους στόχους πολιτικής εντός του μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Με μια συγκριτική αξιολόγηση, θεσμική ανάπτυξη γνώσεως κτλ. Για τους δείκτες, η εποπτεία βασίζεται στο αποκαλούμενο MIP Scoreboard, δηλαδή τους δείκτες που χρησιμοποιούνται για τις διαδικασίες δημοσιονομικής ανισορροπίας που παρέχουν τις βασικές πληροφορίες έγκαιρης, έγκαιρου εντοπισμού δημοσιονομικών αποκλήσεων που μπορεί να εμφανίζονται σε συγκεκριμένες χώρες. Παρακολουθεί ο μηχανισμός λοιπόν τι συμβαίνει στις χώρες και κατά πόσον υπάρχει κίνδυνος σημαντικών δημοσιονομικών προβλημάτων. Αυτός ο βαθμολογικός πίνακας, το scoreboard, είναι πολύ εμφανές και πολύ σημαντικό στην πολιτική συζήτηση, τον πολιτικό διάλογο. Δηλαδή πώς μπορεί να συμπεριληφθεί η απασχόληση και η κοινωνική πολιτική εντός του βαθμολογικού αυτού πίνακα. Στη διαφάνεια αυτή βλέπετε την διαδικασία του εξαμήνου. Πρόκειται για μια περίπλοκη, όπως έλεγα, διαδικασία συντονισμού με διαφορετικά βήματα που καλύπτουν όλο το έτος. Αποκαλείται εξάμεινο γιατί προηγουμένως είχε αυτή τη διάρκεια, τώρα επεκτάθηκε προκειμένου να επιτρέψει πληρέστερη συζήτηση σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο με την συμμετοχή κοινωνικών ενδιαφερομένων φορέων στη συζήτηση και με τη συμμετοχή όλων των ευρωπαϊκών οργανισμών, ιδρυμάτων, κοινωνικών φορέων και, της, και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Περίπλοκη λοιπόν όπως έλεγα διαδικασία την οποία περιγράφουμε λεπτομερώς στη μελέτη δεν θα επεκταθώ σε αυτό γιατί αυτό θα απαιτούσε πολύ χρόνο. Εδώ θα ήθελα να εστιαστώ στα βασικά ζητήματα που απορρέουν από την μελετή. Το πρώτο πόρισμα είναι ότι πλέον αναγνωρίζεται από όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς ότι υπάρχει ανάγκη μεγαλύτερης διείσδυσης της κοινωνικής πολιτικής στο εξάμεινο και καλύτερης ισορροπίας μεταξύ των, μηχανισμών μακροοικονομίας και δημοσιονομικών και των κοινωνικών πολιτικών. Μια καλύτερη ισορροπία δηλαδή μεταξύ των δημοσιονομικών και κοινωνικών προβλημάτων και της αντιμετώπισης τους. Το κέριο ζήτημα είναι πώς θα πρέπει να γίνει αυτό και επ' αυτού συνεχίζεται η συζήτηση. Γιατί είναι πιο σημαντικές πλέον οι ανισορροπίες, διότι οι εμπειρικές ενδείξεις και βιβλιογραφία που έχουμε μας δείχνουν ότι αν δεν εξετάσουμε το ζήτημα απασχόλησης και κοινωνικών προβλημάτων στην οικονομική πολιτική, ο κίνδυνος είναι ότι οι ανισορροπίες που μπορεί να αναπτυχθούν λόγω της ανάληψης των μέτρων λιτότητας θα μπορούσαν να έχουν πολύ σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη και πορεία του μέλλοντος. Υπάρχει μια θετική παράλληλη σχέση μεταξύ της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης και, και του περιορισμού των εισοδηματικών ανισοτήτων. Πρέπει λοιπόν να διατηρούμε υποέλεγχο την απασχόληση και τα κοινωνικά προβλήματα. Και αυτό λόγω του γεγονότος ότι τα προβλήματα στην απασχόληση και στην κοινωνία που μπορούν να απορρέουν από μέτρα λιτότητος και οικονομικά μέτρα μεγεθύνουν τις πιθανότητες οικονομικών κρίσεων, πολιτικής αστάθειας, αποτροπής των επενδύσεων, ή στην παιδεία, στους ανθρώπινους πόρους, στην επιχειρηματικότητα την ίδια. Και υπό τον τρόπο αυτόν περιορίζουν την μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη. Αυτή η εστίαση είναι ιδιαίτερος ε, χρήσιμη σε οικονομικές και υπο τον τροπο αυτων ενώσεις όπως η εστιαση ειναι ιδιαιτερως χρησιμη σε οικονομικες και λέει ο Μιλήτρια. Διότι μια κρίση απασχόλησης μπορεί να μεταλαμπαδευτεί από μια χώρα σε μια άλλη λόγω της οικονομικής εξάρτησης που υπάρχει μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα των χωρών της Ευρωζώνης. Άρα είναι προς το συμφέρον όλων των κρατών μελών να λαμβάνουν υπόψη τους τον αντίκτυπο των μέτρων λιτότητας στις ε, κοινωνικές ε, ανισότητες. Χρειάζεται λοιπόν καλύτερη ισορροπία μεταξύ των μακροοικονομικών και κοινωνικών πολιτικών, αλλά όπως έλεγα, το πρόβλημα είναι πώς θα το πετύχουμε αυτό, πώς θα το καταφέρουμε. Και πώς θα αναπτύξουμε έναν μηχανισμό συντονισμού και διακυβέρνησης που θα διατηρεί αυτήν την ισορροπία μεταξύ των πολιτικών πώς θα επιτύχουμε καλύτερη ενσωμάτωση και καλύτερη συμμετοχή των κοινωνικών φορέων και πώς θα χρησιμοποιήσουμε με καλύτερο τρόπο τους ε, δείκτες ε, απασχόλησης και τους κοινωνικούς δείκτες στα πλαίσια της οικονομικής εποπτείας. Εξετάζοντας τα πέντε πλέον χρόνια της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου από το 11 ως το 15, βρίσκουμε πράγματι ενδείξεις αυξανόμενης προσοχής στα κοινωνικά ζητήματα στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Υπάρχει μια μικρή αύξηση ε, στις συστάσεις για συγκεκριμένες χώρες σε σχέση με συγκεκριμένα κοινωνικά προβλήματα. Υπάρχει μεγαλύτερη προσοχή σε μια προσέγγιση συγκριτικής αξιολόγησης που προτείνει, συστήνει βέλτιστες πρακτικές και σύγκριση μεταξύ των χωρών ώστε να ενθαρρυνθεί η θεσμική γνώση Υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή των κοινωνικών φορέων στη διαδικασία του εξαμήνου. Υπάρχει αυξημένο ρόλο, επί για την ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ απασχόληση στην προπαρασκευή τη εκθέσεως κομισιών και στον ορισμό των συστάσεων αναχώρα. Και αυτό είναι πολύ πρόσφατη εξέλιξη. Είναι από τον κύκλο πολιτικής του 2014. Υπάρχει αυξημένος ρόλος της Επιτροπής ΕΜΚΟ και SPC ή στην ανάπτυξη και εξέταση αυτών των συστάσεων αναχώρα για την αξιολόγηση της επίδοσης των χωρών και για τους δείκτες που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση αυτή. Υπάρχει επίσης μεγαλύτερη συμμετοχή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών μέσω ενός, ε, μιας τριμερού συνόδου για τον μακροοικονομικό διάλογο και πάλι από το 2014 και υπάρχει μια νέα διαδικασία κοινωνικής αξιολόγησης αντικτύπου για τις χώρες των προγραμμάτων που χρησιμοποιήθηκε πρώτα για την Ελλάδα πέρυσι. Πρόκειται για μια εξάντε κοινωνική αξιολόγηση αντικτύπου. Δηλαδή, τα μέτρα που ζητούνται για τις χώρες προγράμματος για να περιοριστεί το δημόσιο χρέος και οι κοινωνικές ανισορροπίες αξιολογούνται εξάντε υπό την κοινωνική έννοια και την έννοια της απασχόλησης. Τα δυνητικά προβλήματα αυτού του χαρακτήρα αξιολογούνται εκ των προτέρων άλλη μια σημαντική εξέλιξη για μια αυξημένη προσοχή στα θέματα αυτά ήταν η ενσωμάτωση της κοινή ε, έκθεσης ε, δικτών απασχόλησης μαζί με τους επικουρικούς δικτές, δηλαδή οι δίκτες μακροοικονομικής εποπτείας συμπεριλαμβάνουν πλέον δίκτες κοινωνικούς και απασχόλησης και αυτό είναι μια σημαντική εξέλιξη διότι σημαίνει ότι σε αυτήν την αξιολόγηση δυνητικών ανισορροπιών δίδεται πλέον προσοχή και στα κοινωνικά ζητήματα. Και το τελευταίο έτος η Κομισιόν εισήγαγε τρεις ακόμα δείκτες απασχόλησης στο MIP που είναι και αυτό πολύ σημαντικό, γιατί αυτοί οι δείκτες επικεφαλίδας είναι οι πιο σημαντικοί για το πρόγραμμα. Και αυτοί θα χρησιμοποιηθούν στο παρόν πρόγραμμα κύκλου, που αφορούν και οι τρεις στην ανεργία. Ωστόσο υπάρχουν κάποιες αρνητικές πτυχές, η διαδικασία αυτή ακόμη είναι μερική δεν έχει ολοκληρωθεί, μακροοικονομική ε, προσέγγιση επικρατεί κατά 60% των ε, συστάσεων ανά κράτος. Υπάρχει επίσης μεγαλύτερη ανελαστικότητα ως προς το σύστημα, υψηλότερη πολιτική ορατότητα της μακροοικονομικής διαδικασίας εποπτείας σε σχέση με τη στρατηγική 2020 θα πρέπει να βρισκόμαστε στη βάση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Αυτό που συμβαίνει πάντως είναι ότι το Ευρωπαϊκό Εξαμήνου αποκτά ορατότητα σε σχέση με, τη με την μακροοικονομική διάσταση, ενώ η στρατηγική Ευρώπη 2020 χάνει έδαφος. Θα γνωρίζετε ασφαλώς και από τις χώρες σας ότι η συζήτηση αφορά περισσότερο μακροοικονομικές ανισορροπίες και όχι άλλα ζητήματα και επίσης κάτι άλλο, όταν οι συστάσεις αναχώρα καλύπτουν θέματα ανεργίας ή κοινωνικά εστιάζονται κυρίως στο κόστος και την αποτελεσματικότητα και την οικονομική βιωσιμότητα παρά στον περιορισμό της ε, φτώχειας των ανισοτήτων. Το βλέπουμε αυτό κυρίως στις συστάσεις για τις μεταρρυθμίσεις, για τη συντάξη, ε, συστήματα για τα φαρμακευτικής περίθαλψης και ούτω καθεξής. Επίσης, ε, στην εξέταση των περιπτώσεων συγκεκριμένων χωρών και μελέτη με σύγκριση ως προς τις κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες ευρωπαϊκές χώρες των συστάσεων με χώρα προκύπτει πως αυτές οι συστάσεις σε ορισμένες περιπτώσεις δεν δίνουν λύσεις στις κύριες προκλήσεις κοινωνικές, προκλήσεις απασχόλησης κλπ. των χωρών και δεν ε, στηρίζουν τις ευάλωτες ομάδες. Μπορεί να εστιάζονται παραδείγματι σε συγκεκριμένες ομάδες στόχο, τους νέους, σε παραδείγμα, 35% των συστάσεων να χώρα φορούν νέους, ενώ άλλοι στόχοι, οι πιο ηλικιωμένοι και οι άνεργοι κτλ. μπορούν να εντοπίζονται, αλλά πολύ λίγα αναφέρονται σε συστάσεις ανά χώρα σε θέματα φίλου των λιγότερο ε, κατηρτισμένων, των μεταναστών. Χαμηλότερες επίσης ε, είναι, χαμηλότερο το ενδιαφέρον σε σχέση με την υλοποίηση των συστάσεων για την αγορά εργασίας και την κάθε χώρα σε σχέση με τις μακροοικονομικές. Ένα από τα προβλήματα είναι ότι συνήθως οι μεταρρυθμίσεις οι κοινωνικές και της αγοράς εργασίας είναι πολύ πιο δυσεφάρμοστες, χρειάζονται περισσότερο χρόνο και φέρνουν αποτελέσματα ύστερα από μακρότερο χρονικό διάστημα. Έτσι είναι δύσκολο να αξιολογηθεί ε, τι έχει πραγματικά υλοποιηθεί σε σχέση με δημοσιονομικά, νομισματικά ή άλλα μακροοικονομικά μέτρα. Αναχώρα. Και παραμένει χαμηλή η χαμηλό ο βαθμό εμπλοκή των κυβερνητικών οργανώσεων και των κοινωνιών των κρατών μελών. Σε πολλέ περιπτώσει, οι επαφές είναι μεταξύ κυβέρνησης και ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, ενώ η κοινωνική εταιρεία, η οργάνωση κοινωνία των πολιτών, το κοινοβούλιο εμπλέκονται σε πολύ περιορισμένο βαθμό στις διαδικασίες αυτές, όπως βλέπουμε στην Ιταλία, παραδείγμα την πατρίδα μου. Ενώ σε άλλες χώρες, όπως χώρες του βορρά της Ευρώπης, Φιλανδία, Φερρυπίν, είναι πολύ πιο σαφή η ανάμειξη στις προσπάθειες αυτές του ε, τομέα της κοινωνίας των πολιτών και των κυβερνητικών οργανώσεων. Οι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών με τους οποίους ήρθαμε εμείς σε επαφή υπεγράμμισαν την ανάγκη για συγκεκριμένες κατευθύνες γραμμές από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να διευκολύνεται η εμπλοκή τους και σε εθνικό επίπεδο η εμπλοκή δηλαδή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των κοινωνικών εταίρων στις συζητήσεις για την οργάνωση για την προετοιμασία των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων. Και Για τους δείκτες τώρα, όπως ανέφερα νωρίτερα, οι δείκτες ε, που περιλαμβάνονται στις MIP, στο ε, πίνακα δηλαδή μακροοικονομικών ανισορροπιών, έχουν μεγάλη σημασία για την ορατότητα των ζητημάτων που καλούνται να αντιμετωπίσουν βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για τον αρμόδιο για τη λήψη αποφάσεων αλλά και για τα μέσα μαζική ενημέρωση. Πρόκειται για δείκτε δηλαδή πάνω στου οποίου συνήθω σχολιάζουν αυτοί που βρίσκονται πάντα στα πρωτοσέλιδα, αυτοί οι δείκτες δηλαδή του πίνακα μακροοικονομικών ανασυνοσορροπιών και γι' αυτό θα πρέπει να βρίσκονται μέσα στον πίνακα αυτοί οι δείκτες και όχι αλλού. Είπα και νωρίτερα ότι υπάρχουν κάποιοι δείκτες, υπάρχουν τέσσερις κύριοι και έξι επικουρικοί δείκτες από τον πίνακα εκ των 40 εν όλο δικτών. Ωστόσο αυτοί που περιλαμβάνονται στον πίνακα δεν καλύπτουν κοινωνικά ζητήματα, αλλά κυρίως ε, συνθήκες ανεργίας ή αγοράς εργασίας. Επίσης δεν είναι ε, αναλυτική σε σχέση με το φύλλο, την ηλικία, εθνικότητα, επίπεδο μόρφωσης. Άρα δεν μπορούν να καταγράψουν στην πληρότητά τους ε, τα περίπλοκα κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα που μας απασχολούν και καλύπτουν επίσης μόνο περιορισμένο αριθμό ε, κοινωνικών ζητημάτων ή ζητημάτων σχετικών με την απασχόληση. Δεν υπάρχουν δείκτες για τη, μόρφωση. Δεν, υπάρχει ζήτημα, δεν υπάρχουν δείκτες σε σχέση με τις ανισότητες ως προς το φύλλο ή την ε, κατάσταση της υγείας. Και έτσι, και για να ολοκληρώνω, με τη μελέτη αυτή εμείς προτείνουμε το εξής. να συμπεριληφθούν νέοι συμπληρωματικοί δείκτες στον πίνακα αποτελεσμάτων MIP, ώστε να είναι πιο ορατή η κίνδυνη ανισορροπιών, ο υπολογισμός των κινδύνων και προτείνουμε δύο νέους δείκτες, κύριους δείκτες, τον κίνδυνο δηλαδή φτώχειας μετά κοινωνική μεταφορά, δεν υπάρχει ένας τουλάχιστον, τουλάχιστον κοινωνικός δείκτης στους κύριους δείκτες, γιατί δεν έχουμε κανέναν αυτή τη στιγμή. Το δε πρόγραμμα σε σχέση με τον δείκτη αυτό είναι ότι είναι ζήτημα το πώς θα υπολογίζεται χώρα και η χρονική στιγμή της καταγραφής. Αυτό το άλλωστε και το επιχείρημα όσων στάθηκαν κατά τη ενσωμάτωση αυτού του δίκτυ στο πίνακα αποτελεσμάτων. Όμω είναι πολύ σημαντικό να, το έχουμε, να τον έχουμε τον δίκτυ αυτό και πρέπει η Eurostat να κάνει προσπάθειες και επενδύσεις για να βελτιώσει το δίκτυ και τη σχετική βέβαια συλλογή δεδομένων ώστε να είναι στο δυνατόν πιο γερά τα στοιχεία πάνω στα οποία θα εδράζεται. Και ο άλλος δείκτης που θέλουμε είναι μακροπρόθεσμο ποσοστό ανεργίας, ε, μάλλον ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας, έτσι ώστε να προβλέπεται ο κίνδυνος ε, να περιέλθει κανείς σε κατάσταση φτώχειας. Πρόκειται για ένα σημαντικό δείκτη για την παρακολούθηση της πολιτικής της αγοράς εργασίας. Και προτείνουμε επίσης την ενσωμάτωση ενώ, ε, νέα νέων, εννέα νέων συμπληρωματικών ή επικουρικών δικτών, σε τομείς που δεν καλύπτουν αυτή τη στιγμή αυτοί οι δείκτες, σε παραδείγματι ποιότητα εργασίας. Συγκεκριμένα ε, συνθήκες ε, συμβατικής σχέσης προσωρινής ή ορισμένου χρόνου, συσχετισμός απασχόλησης με εκπαιδευτικό μορφωτικό επίπεδο, ένα δείκτη παραδείγματι για το μερίδιο επί του ε, πληθυσμού με τριτοβάθμια εκπαίδευση, το ζήτημα της κάλυψης, ε, το ποσοστό καλύψεως από το Εθνικό Σύστημα Υγείας, τα, οι δημογραφικές τάσεις, ε, ε, παραδείγματι ποσοστό εξάρτησης τρίτης ηλικίας, ανισότητες φύλου, δηλαδή μη προσαρμοσμένο κενό στις αμοιβέ μεταξύ ανδρών και γυναικών και άλλοι βέβαια συνήθεις δείκτες όπως ε, μερίδιο εργαζομένων φτωχών και ποσοστό απασχόλησης αναφύλων. Με τους δείκτες αυτούς λοιπόν μπορούμε πιστεύουμε να καλύψουμε πολύ ευρύτερους τομείς πιθανών ανισορροπιών ε, σε σχέση με κοινωνικές ε, τάσεις και τάσεις απασχόλησης. Υπάρχουν και άλλοι δείκτες που θα μπορούσαμε να προσφέρουμε, να προσθέσουμε. Πρέπει όμως να μπουν τρίτη σε σειρά και ίσως και σε κάποιες περιπτώσεις είναι δύσκολο να υπολογιστούν. Για να καταλήξω, θα πάρω ακόμα πέντε λεπτά, για δύο λεπτά, καλώς. Δύο διαφάνειες έχω τους ή άλλους. Ένα κύριο ζήτημα είναι πέραν της εξέτασης των δικτών να βελτιωθούν τα συστήματα διαχείρισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μια πρόταση εδώ για αποκατάσταση των τελικών στόχων της Στρατηγικής Ευρώπη 2020 και συγκεκριμένα την αντίληψη για τους ε, για τις συστάσεις αναχώρα σε ένα ευρύτερο χρονικό πλαίσιο, ώστε να, γίνονται, να εγγράφονται και να γίνονται κατανοητοί και αναγνώσιμοι και οι δείκτες που έχουν να κάνουν με τη μόρφωση, τη δημόσια υγεία και ούτω καθεξής και επίσης αξιολόγηση των κοινωνικών επιπτώσεων, βελτίωση της διαφάνειας και της λογοδοσίας και της ευελιξίας της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου με περισσότερη επικοινωνιακή ε, ε, αντιπαράθεση και ε, δραστηριότητα, ενσωμάτωση, ευελιξία. σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ανταποκριθούν στις κατευθύνες γραμμές και τα ζητήματα πολιτικής ε, που επισημαίνει το ευρωπαϊκό, τα ευρωπαϊκά δεσμικά όργανα για τις χώρες. Και αυτό σημαίνει μια πιο, ένα πιο ήπιο μηχανισμό συντονισμού. αντί για τις πολύ και άτεγκτες μεθόδους ε, της μακροοικονομικής επαγρύπνησης υποπτίας. Και έτσι μπορεί να βελτιωθεί και η αποδοχή της διαδικασίας. Για να κλείσω λοιπόν συγκεκριμένα ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πεδίο αυτό. Βασική ιδέα είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να προσφέρει πολιτική υποστήριξη και περισσότερη εξισορρόπηση μεταξύ πολιτικών στόχων κοινωνική πολιτικής, ιδιαίτερα με την προαγωγή δημόσιου διαλόγου για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και τις συνέπειες που έχουν οι συστάσει αναχώρα σε σχέση με την απασχόληση με τα λοιπά κοινωνικά θέματα και βεβαίω μπορεί το Κοινοβούλιο να υποστηρίξει περισσότερο την συμμετοχή των εθνικών και ευρωπαϊκών εμπλεκομένων φορέων στη διαμόρφωση του εξαμήνου. Παραδείγματι, να γίνονται ακροάσεις, δημόσιος διάλογος για τα ζητήματα του εξαμήνου. Επίσης, μπορεί το Κοινοβούλιο να υποστηρίξει επενδύσεις σε ε, πιο στεναρούς, πιο σωστούς δείκτες κοινωνικού συλλογή δεδομένων, γιατί υπάρχουν δεδομένα που συλλέγονται σε μακρό χρονικό διάστημα και άρα χρειάζονται οι πόροι εκείνοι που θα υποστηρίξουν την συλλογή και προσφορά εξασφάλιση δεδομένων ε, αυτού του χαρακτήρα. Αυτό μπορεί να το προσφέρει ως υποστήριξη λοιπόν στην Επιτροπή και τη Γιούρος από το Κοινοβούλιο. Επίσης αξιολόγηση επιπτώσεων που θα πρέπει να γίνεται σε κάθε πολιτική λιτότητα ε, που θα προτείνεται στις ευρωπαϊκές χώρες και επίσης παρακολούθηση της ε, υλοποίησης των προτάσεων του εξαμήνου. Για να επιτευχθεί λοιπόν ένας πιο σαφής ρόλος, η επίτευξη και των στόχων αυτών. Πιστεύουμε ότι η δημιουργία μια ομάδα εργασία για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο θα ήταν χρήσιμη γιατί θα υποστήριζε έτσι τη συνεργασία μεταξύ τη Επιτροπή Απασχόληση και τη Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με ενίσχυση αντίστοιχα και του ρόλου του Κοινοβουλίου στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και με συγχωρείτε που μακρηγόρησα. Καλώς και σας ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ερωτήσεις ή μήπως και τα επιχειρήματά σας ήταν ενδιαφέροντα. Θα συνεχίσουμε τη συζήτηση όσο έχουμε διαρμηνία κυρία Ιασλοβιέτσκα από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής μας. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σα ευχαριστώ για τις πληροφορίες τις οποίες μας δώσατε. Είναι σαφώς ενδιαφέρουσες, ιδιαίτερα σήμερα όπου βλέπουμε σε βάθος αλλαγές στην αγορά εργασίας. Είπατε ότι μεταξύ των συστάσεων σας Υπάρχει μία η οποία υποστηρίζει ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν περισσότεροι δείκτες για την αξιολόγηση της αγοράς εργασίας. Είπατε επίσης ότι η συλλογή πληροφοριών είναι κάτι το σημαντικό για τον τρόπο που γίνεται. Όταν ακούω ότι στο εσωτερικό της Ένωσης έχουμε δύο εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης χειρεύουσες, διότι δεν υπάρχουν οι κατάλληλοι εργαζόμενοι και από την άλλη έχουμε πάρα πολλά εκατομμύρια ανέργων, διαρωτώ πού είναι το λάθος. Ίσως τα δεδομένα λοιπόν τα οποία συλλέγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συλλέγονται μόνο σε εθνικό επίπεδο, κάτι το οποίο δεν αποδίδει την σωστή κατάσταση της αγοράς. Θα συμφωνήσω μαζί σας, όπου το μίσος τους οποίους καλύπτουν τα εθνικά δεδομένα ε, έχουμε κάποια στοιχεία, αλλά η αγορά εργασίας είναι τόσο ευαίσθητη και όταν οι εθνικές πληροφορίες δεν καλύπτουν το περιφερειακό επίπεδο, τότε πράγματι η προσπάθεια συλλογής των στοιχείων θα πρέπει να γίνει σε τοπικό επίπεδο. Ποια είναι η γνώμη σας γι' αυτό. Κυρία Χάρκιν. Να σας ευχαριστήσω για την έκθεσή σας. Θέλει ξενύχτια πολλά για να μπορέσει κανείς να τα καλύψει όλα αυτά. Να κάνω κάποια σύντομα σχόλια. Εκτιμώ ιδιαίτερως την στάση σας και είναι χρήσιμα τα στοιχεία τα οποία συλλέγεται, ότι δηλαδή οι ανισότητες επηρεάζουν την περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη. Αυτό είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε εδώ και αρκετό καιρό, αλλά το έχουμε αγνοήσει εν πολλής. Πιστεύουμε ότι μόνο η ανάπτυξη θα καλύψει τα προβλήματα απασχόλησης. Ξέρετε ότι στην Ιρλανδία Η παλήρια κανονικά θα πρέπει να ανυψώνει τα πλοία, αλλά αυτό δεν ισχύει στην ουσία, απλά τα κάνει να εξοκύλουν. I think you some very good ideas, but immediately the, Λοιπόν, πολλά από τα στοιχεία λέγουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παρεμβαίνει ιδιαίτερος και δεν έχει τις αρμοδιότητες που απαιτούνται. Αλλά παρόλα αυτά, Περιμένω τις δικές σας απαντήσεις περισσότερο στις παρατήρησεις μου. Τώρα για τους δείκτες, τους κεντρικούς δείκτες και οι κίνδυνοι φτώχειας και οι δυνατότητες που μας δίδουν τα πρόσφατα στοιχεία για τη δική μου χώρα πάντα, ότι πριν από τις κοινωνικές λεγόμενες εσωτερικές μεταφορές, τα επίπεδα ανισότητας ήσαν ήδη ιδιαίτερα ψηλά στην Ευρώπη. Μετά από τις κοινωνικές μεταφορές βρισκόμαστε πάνω κάτω στο μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι πριν από αυτού του επίπεδου τις κοινωνικές μεταφορές τα στοιχεία τα οποία είχαμε ήταν πολύ σημαντικά. Και νομίζω ότι η πρόταση την οποία κάνατε για μια ομάδα εργασίας ανάμεσα στην Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή τη δική μας είναι μια πάρα πολύ καλή ιδέα σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Κάποιοι από εμά είμαστε πλήρη μέλη στη μία Επιτροπή και αναπληρωτές στην άλλη. Είναι μια καλή ε, ιδέα γιατί πώς μπορεί να περιμένει κανείς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να μπορέσουν να διακρίνουν τη σημασία των διαφόρων δικτών αν εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο δεν κάνουμε την σωστή αυτή διάκριση. Μετά την τρίτη ερώτηση μπορείτε να δώσετε απαντήσεις συνολικά. Η κυρία Σόιντροβα. Já děkuji také za e, tuto prezentaci a e, chtěla bych položit otázku, která se... Θα ήθελα να θέσω μία ερώτηση σχετικά με τους δείκτες και σχετικά με την ανισότητα ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες και σε επίπεδο εισοδημάτων και σε επίπεδο συντάξεων. Ξέρετε ότι υπάρχει πάντα μια μεγάλη διαφορά πάντα οι λόγοι για τους οποίους υπάρχει διαφορά διαφοροποιούνται. Μεταξύ των άλλων προβλημάτων είναι η λεγόμενη βοήθεια προς τα παιδιά. Σε ορισμένες χώρες υπάρχουν κάποιες μελέτες, όχι σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά σε εθνικό επίπεδο για την κατάσταση αυτή. Δεν θα μπορούσαμε να προβλέψουμε ένα νέο δίκτυο, ο οποίος να κάνει τη διάκριση ανάμεσα στα εισοδήματα των ανδρών και των γυναικών που ασχολούνται με τα παιδιά τους γιατί τέτοιου είδους δείκτες δεν υπάρχουν. Θα ήταν ένας δείκτης ο οποίος θα ήταν πάρα πολύ πιο χρήσιμος έτσι ώστε να διακρίνουμε την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα παιδιά που φροντίζονται από τους γονείς τους και τα παιδιά τα οποία σε κάποια φάση μπαίνουν στην αγορά εργασίας και αλλάζει η κατάστασή τους και σε επίπεδο μισθολογικό. Λοιπόν, κυρία Λοντοβίτσι, Αυτές είναι ερωτήσεις που είχα να σας θέσω. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Πράγματι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία η ανάλυση των στοιχείων σε περιφερειακό επίπεδο. Χρειαζόμαστε τα περιφερειακά στοιχεία διότι οι διαφορές είναι πάρα πολύ μεγάλες. Εγώ προέρχομαι από μια χώρα και το θέμα των διαφορών ανάμεσα στον Βορρά και τον Νότο είναι καθοριστικό. ανάμεσα στους ε, εμπλεκομένους που πήραμε συνεντεύξεις, ε, πολλοί έθεσαν το θέμα των διαφορών των περιφερειακών και ασκήθηκε κριτική στις συστάσεις αναχώρα, διότι δεν έλαβαν υπόψη τις περιφερειακές διαφορές. Συνεπώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούσε να προωθήσει να υπάρξει μεγαλύτερη χρήση των περιφερειακών δεκτών. Ε, βελτιώνονται. Εγώ άρχισα να ασχολούμαι με τα θέματα αυτά τα περιφερειακά εδώ και 20 χρόνια και δεν υπήρχε τίποτα. Τώρα έχει υπάρξει ένας περιφερειακός δείκτης που έχει πολλούς επιμέρους δείκτες αλλά δεν αρκεί. Σας ευχαριστώ λοιπόν για τον συσχετισμό της ανισότητας από τη μία και της ανάπτυξης από την άλλη. Είναι προφανές ότι η ανισότητα μπορεί να επηρεάζει την ανάπτυξη. Ενώ δεν είναι ξεκάθαρο το εάν η υψηλότερη ανάπτυξη σημαίνει και υψηλότερη ισότητα. Υπάρχει το γνωστό βιβλίο του Πικετή, το κεφάλαιο, χίλιες σχεδόν σελίδες, που αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει θετικός συσχετισμός ανάμεσα στην οικονομική ανάπτυξη από τη μία και την ισότητα ή καταπολέμηση της ανισότητας από την άλλη. Εξαρτάται λοιπόν από τις πολιτικές οι οποίες ακολουθούνται στις φάσεις της ανάπτυξης και οι οποίες επιδιώκονται και εφαρμόζονται από τα κράτη. Τώρα για τις εθνικές αρμοδιότητες και τις κοινοτικές αρμοδιότητες. Αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο τα θεσμικά όργανα της Ένωσης απέκτησαν θα έλεγα μεγαλύτερες εξουσίες, αρμοδιότητες για να μπορούν να κάνουν α, συστάσεις όχι μόνο για την Ευρωζώνη, για τις χώρες της Ευρωζώνης αλλά και για κοινωνικά θέματα. Συνεπώς υπάρχει μια κάποια συζήτηση στην παρούσα φάση ανάμεσα στα κράτη-μέλη και τα ευρωπαϊκά όργανα. Μία από τις ε, αντιφάσεις που υπήρχαν σε σχέση με τη χρήση, αντιθέσεις μάλλον, με τη χρήση επιπλέον δικτών κοινωνικών στο ε, πίνακα MIP, στο, σχετικά με το εσωτερικό ακαθάριστο, ε, οφείλεται στο ότι οι δείκτες θα πρέπει να ε, καλύπτουν ένα συγκεκριμένο χώρο και στον τομέα των κοινωνικών. Και γι' αυτό η διεύρυνση των δικτών δεν θεωρήθηκε σωστή. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο πιστεύουμε εμείς ότι η ανοιχτή μέθοδος συνεργασίας είναι ένας σωστός τρόπος συνεργασίας του θέματος των αρμοδιοτήτων. ιδιαίτερα όταν μιλάμε για τα θέματα της απασχόλησης και τα κοινωνικά θέματα, τα οποία εξαρτώνται πολύ από τις τοπικές συνθήκες. Σχετικά με τους δείκτες, εμείς θεωρούμε ότι μετά από τις κοινωνικές μεταφορές υπάρχουν κίνδυνοι στον κοινωνικό τομέα. Εμείς τους δείκτες αυτούς τους χρησιμοποιούμε μετά τις κοινωνικές επαναλαμβάνω μεταφορές, έτσι ώστε να έχουμε κάποιες τάσεις για τον ρόλο των κοινωνικών πολιτικών και της πιθανής μείωσης ε, των κινδύνων για τη φτώχεια. Έτσι θα μπορέσουμε να κρίνουμε πώς οι χώρες μπορούν να μειώσουν την ανισότητα μέσω των κοινωνικών εταίρων, μέσω των κοινωνικών πολιτικών και η Ιρλανδία είναι ένα καλό παράδειγμα πολιτικών που μπορούν να βοηθήσουν τους κινδύνους για τη φτώχεια. Η Ιταλία είναι στην αντίθετη κατάσταση. Δεν έχουμε καλές πολιτικές για τη μείωση των κινδύνων. Συνεπώς η, χρήση, η σύγκριση που κάνετε ήταν μια χρήσιμη σύγκριση. Τώρα για την ομάδα εργασίας του εξαμήνου χαίρομαι που μπορεί να θεωρηθεί χρήσιμη για τις ανισότητες σε επίπεδο φύλων φυσικά για να εξηγήσουμε τις ανισότητες που οφείλονται στη διαφορά των φύλων υπάρχουν πολλοί παράγοντες και ένας από τους πιο σημαντικούς είναι η δυνατότητα φροντίδας για τα παιδιά, ηλικιωμένους, αναπήρους κτλ. Το πρόβλημα με την επιλογή των δικτών είναι ότι έχουμε ένα πλήρη κατάλογο σχετικά με τα ποσοστά κάλυψης της φροντίδας των παιδιών. Έχουμε το στόχο της Βαρκελόνης κατά 30%. Υπάρχει δείκτης που χρησιμοποιείται δηλαδή από τη Eurostat, αλλά δεν έχει προταθεί ε, στον μικρό κατάλογο των δικτών, γιατί όπως ξέρετε δεν μπορούμε να έχουμε πάρα πολλούς δείκτες. Η βασική ιδέα είναι να χρησιμοποιήσουμε ένα μικρό κατάλογο δικτών που μπορεί να ισχύσει για όλες τις χώρες και ίσως θα μπορούσε να υπάρξει ε, ένας διαφορετικός κατάλογος πολύ ευρύτερο σε μια ιστερότερη φάση με πολύ περισσότερους δείκτες. Σας ευχαριστώ λοιπόν για τα σχόλιά σας. And thank you. Και εμείς σας ευχαριστούμε λέει η Πρόεδρος που ήσασταν εδώ μαζί, μαζί μας σήμερα παρότι δεν είμαστε και πολλοί στην αίθουσα όπως βλέπω. αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που μας παρακολουθούν από το δίκτυο μπροστά στον υπολογιστή τους. Είναι όμως ένα από τα βασικά ζητήματα με τα οποία ασχολείται η Επιτροπή μας. Σας ευχαριστούμε για την παρουσίαση, για τη μελέτη και για την παρουσία σας εδώ. Το οποίο μας οδηγεί στην ολοκλήρωση της πρωινής συνεδριάσεως. Θα τα ξαναπούμε στις 3 το απόγευμα και θα ξεκινήσουμε με την ψηφοφορία. Φροντίστε παρακαλώ να είστε εδώ. Μετά την ψηφοφορία έχουμε λιγότερο ενδιαφέροντα πράγματα να ακούσουμε. Ευχαριστώ προς το παρόν.